Καλησπέρα σε όλους. Μπορούμε να αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Ξεκινάμε. Είναι δύο μέρες πολύ σημαντικές για την Επιτροπή μας. Ξεκινάμε με μία μικρή τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Αφορά στη συνεδρίαση αύριο το απόγευμα. Θα ήθελα να αλλάξουμε τα σημεία 11 και 12. Το, το 12 γίνεται 11 για την κατάσταση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων πριν από την έκθεση του Μάρτιν Χάουσλινγκ για την βιολογική παραγωγή. Και αν δεν έχετε παρατηρήσεις γίνεται αυτή η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη για αύριο το απόγευμα. Για τεχνικούς λόγους έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα λιθουανικά και ζητούμε συγγνώμη. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών της 23ης-24ης Απριλίου του 12 και συνεδρίαση της, ε, πρακτικά της 8ης Μαΐου του 12. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται, αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο σήμερα. Ξεκινάμε με το σημείο 4. Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων. Κανονισμός ενιαίας κόρ. Ο Μισελ Νταντέν είναι ο εισηγητής, οι σκιώδεις εισηγητές είναι παρόντες και θα τους δώσω το λόγο μετά τον Μισελ. Ξεκινάμε, συνάδελφοι, ξεκινάμε μια πολύ σημαντική φάση των νομοθετικών εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ με την παρουσίαση των εισηγήσεων για τις τέσσερις βασικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση άμεσες πληρωμές, ανάπτυξη της υπαίθρου, ΚΟΑ και οριζόντιος κανονισμός. Εμείς σήμερα ξεκινάμε με την ενιαία ΚΟΑ και ο Μισελ Νταντά είναι εισηγητής. 10 Ιουλίου λήγουν οι προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψη όμως και τον τεράστιο όγκο των ντοσιέ για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ, τυπωμένο χαρτί δηλαδή, σας παρακαλώ να κρατάτε τα αντίγραφά σας για τις επόμενες συνεδριάσεις. Δεν θα ξανατυπωθούν. Ευχαριστώ και τον Διευθυντή Πατσέκο που είναι παρόν και δίνω το λόγο στον Μισελ Νταντάν για την παρουσίαση. Μισελ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ενιαία ΚΟΑ είναι ένα κείμενο μακροσκελές και σύνθετο από νομικής και νομικής ε, πλευράς, είναι όμως ένα θεμελιώδες κείμενο για την ΚΑΠΑ. Θα ήθελα, πλην παρουσιάσω την έκθεσή μου, να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με βοήθησαν στην δουλειά μου. Σε μεγάλο βαθμό μέσω αυτού του κανονισμού ορίζουμε το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται η γεωργία και η αγροτροφημική βιομηχανία της Ένωσης. Μέσα από αυτόν τον κανονισμό αναπτύσσουμε το όραμά μας για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Χωρίς εμείς να αλλάξουμε ριζικά την αρχική πρόταση της Κομισιόν, θέλησα να ορίσω μερικές ισχυρές πολιτικές θέσεις και να ορίσω και μια πλατφόρμα σκέψης που θα πρέπει να εμβαθύνουμε μαζί. Ο πρώτος άξονας που θέλησα να εμβαθύνω είναι η ασφάλεια και η οικονομική ορατότητα των παραγωγών και των δικτύων παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ιδιώτες να έχουν σαφείς κανόνες για το πώς ρυθμίζονται οι αγορές. Κανόνες που δεν θα είναι αμφίβολοι ως προς την ερμηνεία. Η δημόσια παρέμβαση και η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθήκευση θα πρέπει να ξεκινούν αυτόματα όταν έχουμε τα κατόφλια, τα κατε, κατεπήγοντα. Δεν πρέπει δηλαδή η Κομισιόν να αντιμετωπίσει όπως την κρίση του γάλακτος το 2008-2009 να την αφήσουμε έτσι και να δημιουργήσουμε και σύγχυση σε ήδη τεταμένες αγορές. Προτείνω λοιπόν η τιμή αναφοράς να αναλαμβάνει υπόψη της την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, του κόστους των εσόδων και της εξέλιξης της αγοράς. Εγώ θα ήθελα να γίνει και μία σαφής εξήγηση για το περιθώριο κέρδους των παραγωγών για το βόλιο κρέας να ανέλθει στο 80% της τιμής αναφοράς να πάμε στα, στις 2.000 ευρώ τον τόνο πράγμα το οποίο να, το τη φέρει στο επίπεδο της αγοράς βάσει της τιμής αναφοράς. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα διότι η τιμή παρέμβασης και η τιμή αναφοράς στο βόλιο κρέας είναι ο μόνος, ο μόνος τομέας όπου δεν υπάρχει αλληλοσύνθεση για το ελαιόλοδο, τιμή αναφοράς. Για το έξτρα παρθένο αυξάνω τις τιμές και ζητώ από τον κλάδο να βελτιώσει την ποιότητα. Για τα επιλέξιμα προϊόντα στους δύο μηχανισμούς θέλω στην, ε, στον κατάλογο για το ιδιωτικό για την ιδιωτική αποθήκευση να μπουν τα τυριά, το κατσικίσιο κρέας, οι ελιές κλπ. Επίσης, προτείνω έκτακτα μέτρα συνολικά για το παράρτημα 24, για το 24 του παραρτήματος 1 που θα πρέπει να ενταχθούν στην ΚΟΑ. Χρειάζεται παρακολούθηση της αγοράς, όταν μιλάμε εμείς ότι χρειάζεται δίκτυο προστασίας, κάτι τέτοιο εννοούμε, και οι οικονομικοί χρήστες και η παραγωγή θα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη της ρύθμισης έχοντας πιο εύκαμπτα διαχειριστικά μέσα και αποκεντρωμένα. Οι οργανώσεις των παραγωγών θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των δημοσίων δικήσεων. Θέλω να ενισχυθεί η θέση της Κομισιόν για την ενίσχυση των αγορών των παραγωγών που θα πρέπει να συνενώνονται σε υποδομές με ένα εύλογο μέγεθος για την αγορά. Οι ενώσεις των παραγωγών θα πρέπει να, γίνουν, να μεγαλώνουν για να μπορούν να υπησέρχονται στις αγορές. Το 106 παράγραφος Γ λέει το κείμενο ότι θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός της παραγωγής και προσαρμογή στη ζήτηση και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ρύθμιση απριορή με τη διαχείριση των όγκων και εκ των υστέρων με απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Η προπτική τώρα για την κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος είναι πλέον κοντινή και πρέπει να εξετάσουμε τον τομέα του γάλακτος το πακέτο γάλακτος το οποίο ψηφίσαμε στην αρχή του χρόνου να αρχίσει να εφαρμόζεται, όπως επίσης να φανταστούμε και τον μηχανισμό κρίσης που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιοχές εκείνες όπου αυτή η παραγωγή είναι κυρίαρχη. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω μεγαλύτερη συλλογική και ατομική ευθύνη των διαφόρων παραγωγών. Θα έπρεπε λοιπόν η Κομισιόν να ενισχύσει τους παραγωγούς εκείνους που μειώνουν κατά 5% την παραγωγή γάλακτος έναντι της προηγούμενης χρονιάς και αυτό σε μια προθεσμία τριών μηνών. Το γάλα το οποίο χορηγείται δωρεάν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις επίσης θα πρέπει να αφαιρείται. Θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόστιμα αυτοί οι οποίοι αυξάνουν την παραγωγή στην ίδια περίοδο και κατά την ίδια αναλογία. Όταν θα έχουμε λοιπόν όσοι μάλλον δεν ξεπερνάνε αυτό το όριο της, ε, του 5% στην περίοδο της κρίσης δεν θα πρέπει να τιμωρούνται. Για την ασφάλεια και για την ορατότητα των οικονομικών χρηστών θα πρέπει να έχουμε και έναν άξονα που θα ενισχύει την οργάνωση κλάδου μέσα από την ενιακόα με αύξηση των δυνατοτήτων των παραγωγών. Ξέρουμε όμως ότι η ΚΑΠ στο μεταξύ έχει αλλάξει. Ξέρουμε ότι έχουν αποδυναμωθεί οι παραγωγοί με μείωση του εισοδήματός τους. Θα πρέπει να τους ενισχύσουμε συσπυρώνοντάς τους και αυτό αποτελεί βασική αρμοδιότητα για την ΚΟΑ. Δεν θα πρέπει βέβαια να δημιουργηθούν καρτέλ τα οποία δεν θα βοηθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών. Αλλά θα τους επιτρέψει αυτή η συσπήρωση, αυτή η συνένωση να ξεφύγουν από την οικονομική εξάρτηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους καταναλωτές. Η πολιτική των χαμηλών τιμών έχει ένα αντιστάθμισμα και κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό. Χρειάζεται μία χρυσή τομή για την αηφόρο ανάπτυξη. Θα ήθελα να διαγραφεί εκείνη η ρήτρα που λέει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση της δεσπόζουσας θέσης από τις ενώσεις των αγροτών. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η δεσπόζουσα θέση, η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης καταδικάζεται από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Όταν ε, μία, ένα συνεταιρισμό παραγωγών ε, καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση σημαίνει ότι έχει πετύχει και μεγαλώνει. Το νέο περιθώριο χειρισμών θα πρέπει να συγκεντρώνεται στην καινοτομία, στην πρόληψη και στη διαχείριση των κινδύνων Όπως επίσης ε, Όπως επίσης η παραγωγή του κλάδου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται άμεσα με τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους τα συμβόλαια τους. Θα πρέπει να επιτρέψουμε το συνεταιρίζεστε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες για τις κοινέ δράσεις. Πρώτο δίκτυο ασφαλείας για τον παραγωγό είναι οι τιμές της αγοράς. Είναι θεμελιώδες λοιπόν αυτή η λογική να περνάει μέσα από την κοινή δράση και να βασίζεται στη βασική εμπορική πράξη, στη διαπραγμάτευση ενός συμβολέου με μία τιμή. Προτείνω κατά συνέπεια τη λογική του πακέτου γάλακτος να την επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα πακέτα. Διάλογο μεταξύ γεωργικών κλάδων και γεωργικοτροφημικής βιομηχανίας, διαπαγγελματικός διάλογος σε όλους τους τομείς, με διευρυμένες αρμοδιότητες έναντι της πρότασης Κομισιόν, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να υποκαταστήσουμε αυτήν την κουλτούρα συνεργασίας, να, να, τους προτρέψουμε προς μια κουλτούρα συνεργασίας αντί της υψίουσας κουλτούρας αντιπαράθεσης. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικό και για τους καταναλωτές. Πέρα λοιπόν από τους ρόλους που έχουν αναλυφθεί στις, ε, από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών θα ήθελα να λάβουν υπόψη τους και το θέμα του κόστους παραγωγής και της τιμής να έχουν πρόβλεψη της ε, παραγωγής και διαπίστωση των τιμών αγοράς και νοτομία και εφαρμογή συλλογικών διαβημάτων τα οποία θα μας προφυλάσσουν από φυτο ε, και περιβαλλοντικούς κινδύνους όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τώρα, για την συμβολή, την χρηματική συμβολή των διαφόρων μελών σε αυτές τις ε, επαγγελματικέ οργανώσεις δεν αλλάζω τίποτα στην οργάνωση που προτείνει η Κομισιόν. Πρόκειται για κυβερνητικές αποφάσεις, οπότε τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να αποφασίσουν. Δεν πρόκειται για ιδιωτικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στη δράση των διαφόρων γεωργικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, έτσι όπως ορίζονται από τα άρθρα 106-108 καλύπτονται όλα τα προϊόντα τα οποία είναι εμπορεύσιμα στα κράτη-μέλη αλλά και τα εισαγόμενα τα οποία θα συμμετείχαν σε συλλογικές ε, ε, δράσεις όπως είναι οι διαφημιστικές ε, εκστρατείες. Θα πρέπει να προβλέψουμε επίσης τη διαφάνεια της αγοράς για να διαφωτίσουμε και τους οικονομικούς χρήστες και όλους τους ενδιαφερόμενους το 116α προτείνω να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου παρακολούθησης των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Και αυτός ο νέος οργανισμός θα πρέπει να δημιουργηθεί στα πλαίσια της Eurostat. <coughs> Για να έχουμε όμως πραγματικές εξελίξεις επί τόπου, χρειάζεται οι οργανώσεις των παραγωγών να λειτουργούν εύρυθμα, να μπορούν να υπάρχει σαφής κώδικας για τον ανταγωνισμό ο οποίος να τηρείται. Στο λέγεται ότι οι κανόνες για τον ανταγωνισμό δεν θα πρέπει να εμφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα έτσι, παρά μόνο όταν ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτός ο όρος δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από την Ρώμη και μετά, αλλά δεν εφαρμόστηκε και ποτέ. Στο τέλος είναι. Από το 60 και μετά δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα. Εκπλήσωμε όταν η Κομισιόν προτείνει αυτό το νέο πλαίσιο ανταγωνισμού για τις γεωργικές δραστηριότητες, αγνοεί αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν επικαλείται τις νομικές βάσεις. Στο παρελθόν αυτά τα μέτρα για τον ανταγωνισμό ίσχυαν διότι υπήρχε μεγάλη κρατική παρέμβαση στον τομέα της ε, γεωργίας, αλλά με τις μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να αλλάξουμε. Έτσι όπως έχουν αλλάξει σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να έχουμε μία αντιμετώπιση σχετικά παρεκκλητική από τον κώδικα του ανταγωνισμού. Επιπλέον, η εφαρμογή του δικαίου για τον ανταγωνισμό είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα με διαφορετικές ερμηνείες και με εντελώ διαφορετικές δράσεις μεταξύ των κρατών μελών. Είναι θεμελιώδες από τώρα να έχουμε συζήτηση για αυτό το ζήτημα για το οποίο οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές στην εσωτερική αγορά. Αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια νέα ερμηνεία των κανόνων του ανταγωνισμού όπως επίσης να ορίζεται η δεσπόζουσα θέση εν μέρη ως βαθμός συγκέντρωσης αποδεκτός σε έναν τομέα Και εγώ λοιπόν πρότεινα σημεία προς ε, σκέψη και, και ανάλυση. Εγώ ελπίζω σήμερα να έχω προτάσεις ε, βελτίωση στο κείμενο. Επίσης θεώρησα σημαντικό να ξεκαθαρίσω το κείμενο της Κομισιόν σχετικά με την εξέρεξη στο δικαίωμα του ανταγωνισμού. Όσον αφορά στις οργανώσεις των παραγωγών πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η προϋπόθεση συμβατότητας των συμφωνιών συμφωνίες ε, και διαβουλευμένες πρακτικές μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών με τους στόχους ε, της ε, ΚΑΠ, έτσι όπως εξαντέρνονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης. Μία συχνή νομολογία θεωρεί ότι για να θεωρείται απαραίτητο για τους, ότι πληρεί τους στόχους της συνθήκης και ότι είναι συμβατό με τους κανόνες ε, του ανταγωνισμού, οι συλλογικές πρακτικές των οργανώσεων των παραγωγών θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση συνολικά των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου και όταν αυτές είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να είναι ένας μεγάλος νομικός για να καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να υπάρχει μια γενική προϋπόθεση συμβατότητας με τους στόχους της ΚΑΠ για τι συμφωνίε που αφορούν στην παραγωγή, την εμπορευματοποίηση, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή την μεταποίηση. Πρόκειται για κάτι το αντίστοιχο με τους υπάρχοντες κανονισμούς που σε άλλους οικονομικούς τομείς δίνουν ε, αμπλοκ ε, ε, εξαιρέσεις, απαλλαγές για ορισμένες οριζόντιες συμφωνίες. Επίσης, ο πρώτος άξονας ασφάλειας και ορατότητας για τους οικονομικούς χρήστες συμπληρώνεται με την με, με τη θετική λίστα των ε, συμφωνιών που εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 101. Επίσης χρειάζεται γράμμιση των διαδικασιών με αυτές που εφαρμόζονται με τους άλλους οικονομικούς τομείς, εφαρμόζοντας το άρθρο, τον κανονισμό, συγγνώμη, ανακάθετος 2003 και η, αρμόδια αρχή είναι αυτή που θα πρέπει να αποδείξει την απαλλαγή από τις ε, ε, από, το δίκαιο του ανταγωνισμού για τις συμφωνίες κλπ. Ε, επίσης, προτείνω σε περίπτωση κρίσης, υγειονομικής κρίσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να υφίσταται ο έλεγχος της Κομισιόν και των κρατών μελών για να ενισχύσουν τον τομέα και να αποφύγει την πτώχευση. Για το γάλα, για το κρασί και για τη ζάχαρη, κρατιέμαι σε αυτά που είπε ο Άλμπερντες τον Ιούνιο. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου έλεγε ότι θα πρέπει ότι έχουμε μέσα σταθεροποίηση της αγοράς επαρκή για την περίοδο μετά το 2015. Για το κρασί και για τη ζάχαρη, σύμφωνο με τη θέση του Κοινοβουλίου που θέλει παράταση του καθεστώς για τις ζαχροχομικές ποσοστώσεις μέχρι το 2020 και τη διατήρηση του καθεστώτος για τα δικαιώματα φύτευσης. Όμως θεωρώ για τον τομέα της ζάχαρης να μπει το βασικό κείμενο ένας μηχανισμός ε, που έχει χρησιμοποιήσει η Δικομισιόν σε μια βάση ad hoc και που επιτρέπει να επανεντάξει στο σύστημα των ποσοστώσεων το σύστημα το, τη ζάχαρη που είναι υποποσοστοτική όταν υπάρχει ανάγκη και έλλειψη. Ένα εύκαμπτο νομικό σύστημα θα επιτρέπει στην Κομισιόν να δρά πιο γρήγορα από ό,τι σήμερα. Τώρα για, το, για τη ζάχαρη διαπίστωσα πόσο ε, διαφέρουν ριζικά οι θέσεις των διαφόρων χρηστών. Μέχρι τώρα δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν να προσεγγίσουν αυτές τις θέσεις. Θα ήταν καλό για όλους στους επόμενους μήνες να βγούμε από αυτές τις ε, στήρες θέσεις και να βρούμε μία θέση <coughs> συνενετική. Για το καθεστώς ενίσχυσης ε, φρούτα και λαχανικά στο σχολείο, γάλα στο σχολείο, προγράμματα εργασίας για τον ε, τομέα του ελαιολάδου και την μελισσοκομεία. Θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινίσουμε το κείμενο της Κομισιόν με τροπολογίες που αφορούν στη γενική φιλοσοφία που ενέκρινε η, Κομισιόν όταν η Επιτροπή μας συγγνώμη, όταν ψήφισε την έκθεση Δεκάστρο για την ε, πρόταση ευθυγράμμισης των ΚΟΑ στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και συμπεριέλαβα την έκθεση Δεκάστρο στη δική μου. Για τα φρούτα και τα λαχανικά προωθούμε την οργάνωση των όπορο-παραγωγών για να μπορέσουν να έχουν ένα μέγεθος ε, επαρκές για να αντιμετωπίσουν τον αγωνισμό και την αγορά στα οποροκυπευτικά. Αυτό προβλέποντας και οικονομικά κίνητρα για την διαχείριση από ενώσεις των παραγωγών αυτών των λειτουργικών προγραμμάτων για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των κρίσεων. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση για την Επιτροπή μας. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο αφορά στο όραμά μας ε, για την μελλοντική ΚΑΠ. Ξέρουμε όμως πως οι θέσεις μας και οι προτεραιότητές μας μπορούν να διαφέρουν σε πολλά. η διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πακέτο γάλακτος απέδειξαν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αυτές όμως οι διαπραγματεύσεις απέδειξαν ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε ευρύτερα σε πολιτικές γραμμές και για σημαντικά θέματα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καρποφόρες συνθήκες για διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Με αντίστοιχο πνεύμα περιμένω τη συνεισφορά σας σήμερα με νέο πνεύμα για να βελτιώσω τις διατάξεις τις οποίες προτείνω στην έκθεσή μου και ούτω ώστε η ΚΟΑ να γίνει πιο αποτελεσματική για να ανταποκριθεί στους στόχους της ΚΑΠ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλη την ομάδα που με βοήθησε, το προσωπικό της Επιτροπής ε, Γεωργίας, την Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, τον Επίτροπο Τσόλους για τις υπηρεσίες του και τον βοηθό μου τον Τενίκη Γέρμη και συγγνώμη από τους διερμηνείς εάν μίλησα γρήγορα. Μπράβο Μισελ, έκανες πολύ σημαντική δουλειά. Μπορούμε να σε ευγνωμονούμε, γιατί είναι πάρα πολύ πλοκό αυτό το ντοσχέ και από νομικής πλευράς και ως προς το όραμα που θέλει να προτείνει για μια νέα κόα. Ευχαριστώ Μισελ. Ξεκινάμε τη συζήτηση, έχουν εγγραφεί όλοι. Να διαχειριστούμε λοιπόν σωστά το χρόνο μας. Να ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Και δίνω το λόγο στην Ιράτσε Γκαρθία Πέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να συμμετέχουν όλοι. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Νταντέν, τον συγχαίρω για τη δουλειά του. Γιατί αυτούς τους τελευταίους μήνες συζήτησης συγκλίναμε πολλοί συνάδελφοι σε αυτές τις βασικές πτυχές ε, που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του εισηγητή. Έχουμε απόλυτη συνείδηση για το πόσο σημαντική είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, για το πόσο είναι σημαντικός ο κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις και την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλλά επίσης έχουμε συνείδηση ότι αν έχουμε και πραγματικά μέσα για τη σωστή πληρωμή των γεωργών ε, καταφέρνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα κείμενο φιλόδοξο και σύμβατο με προηγούμενες ε, θέσεις που έχουν εκφραστεί για τον ανταγωνισμό στο γεωργικό τομέα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ παρουσίασα ως τροπολογία για το γάλα και θεωρώ θεμελιώδες. Είναι η δυνατότητα οι, εθνικές, οι αρμόδιες εθνικές αρχές να συνοντονίζονται ούτω ώστε να έχουν ένα ενιαίο αποτέλεσμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται σήμερα. Εμείς ε, βλέπουμε ότι οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με το κράτος μέλος. Χρειάζεται, είναι θεμελιώδης <coughs> αυτός ο συντονισμός. Ε, οι θέσεις ε, για τις διακλαδικές οργανώσεις, για τους συνεταιρισμούς έχουν ενταχθεί πολύ καλά στο κείμενο. Μετά υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Εγώ μόνο ήθελα να αναφερθώ σε μερικά συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η τιμή αναφοράς ρυζιού πρέπει να αλλάξει, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει αλλάξει και θα πρέπει να έχουμε μια γενική διαδικασία που θα επιτρέπει την αναθεώρηση των τιμών αναφοράς. Στην έκθεση του κυρίου, ο κύριος Νταντέν εναρμονίζει τις ε, καμπάνιες ε, εμπορευματοποίηση, ε, της περιόδους εμπορευματοποίησης των προκυπευτικών με τις περιόδους καλλιέργειας, περιόδους παραγωγής, συγγνώμη. Αλλά η Κομισιόν ήδη το έχει κάνει και ζητάει την εναρμόνιση. Γιατί το διάγραψε ο κύριος Νταντέν για την 93 για το ελαιόλαδο. Εσείς, ε, εσύ, εσείς ε, ε, μιλάτε για το αγνό παρθένο ελαιόλαδο αλλά η αγορά ρυθμίζεται κυρίως από το παρθένο και από το βιομηχανικό ελαιόλαδο. Το απλό ελαιόλαδο. Τώρα για τον αυτόματο, ε, για την αυτόματη τιμή ε, προσαρμογής ε, θα γίνει όπως θα γίνεται με το βούτυρο όπως γίνεται με το βούτυρο επίσης και για τα πουλερικά με το κρέας των πουλερικών θα έχουμε φυγράμιση με εκείνο των κουνελιών τώρα τι να πω για τα προϊόντα κάποιο μπορεί να μας ξεφύγει αλλά μήπως μπορούμε να έχουμε έναν μηχανισμό να έχουμε μια νομική βάση ούτω ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε όταν ένας ε, κλάδος έχει ανάγκη για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός παρέμβασης. Όπως ήδη είπα και μια άλλη φορά, δεν καταλαβαίνω γιατί από τον κανονισμό εξαφανίστηκαν τα ζητούμενα και τα αιτήματα των μεταποιημένων οποροκυπευτικών. Τώρα στην ΚΟΑ λόγω του στην ΚΟΑ είπαμε να μην μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα δεδομένου ότι πρόκειται για μια οριζόντια οδηγία. Αλλά είδα ότι μιλάμε τελικά για το κρασί, για τη ζάχαρη. Ε, γιατί να μην μιλάμε και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Εγώ θα κάνω μια σχετική τροπολογία για να διαγραφούν και αυτά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για, τα, για τις άειλες υπηρεσίες ε, όπως είναι το μάρκετινγκ και να μπορέσουν και, αυτά να, να ενταχθούν ε, μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για την ΚΟΑ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εισαγωγή των κανόνων ε, για τα γαλακτοκομικά. Τον ευχαριστώ και για την παράταση για τη ζάχαρη μέχρι το 2015 όπως και για την ενίσχυση του αμπελικού τομέα. Ξέρω ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ε, απόψεις εδώ μεταξύ των συναδέλφων αλλά πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν στη γραμμή που εγκρίναμε στο παρελθόν και όπου ο κύριος Νταντέν ενέταξε ε, στο κείμενο. Τώρα, επειδή είναι παρούσα η Κομισιόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το συγκεκριμένο στην Κομισιόν. Για τα standard marketing φαίνεται ότι η Κομισιόν τα μετέφερε στην πρόταση για την νέα ΚΟΑ αλλά πάλι για τα οποροκυπευτικά, αυτά που τα οποία τροποποιούν στο 113α το άρθρο 2, ε, τα έχουμε βγάλει από την πρόταση. Αυτό για ποιο λόγο χρειάζεται εξήγηση ή απλώς είναι μία απλή αμέλεια και παραδρομή. Μπορεί η Κομισιόν να μας απαντήσει σχετικά. Ευχαριστώ τον κύριο Νταντέν και όλους όσους ε, συνεργάστηκαν σε αυτή την τόσο την τεχνική έκθεση. Ωραία. Ευχαριστώ Ιράτσε. να καλωσορίσω τον Ερή Κανριέ, ο οποίος αντικαθιστά τον Στεφάν Λαφόλ, ο οποίος από σήμερα είναι ο νέος Υπουργός Γεωργίας στη Γαλλία. Καλώσόρισε, Ερίκ. Η Ρίτα Ρέμερς και μετά ο Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την περιεκτικότατη έκθεσή του, για την περιεκτικότατη παρουσίαση έστω και αν αναφερθήκαμε βιαστικά και δεν ε, εμβαθύναμε και δεν κατάφεραν οι διερμηνείς να ε, εμβαθυνούν και εκείνοι. Έχω ορισμένες ερωτήσεις. Μετά την πρόταση για τις παρεμβάσεις και τους ε, αυτοματισμούς, μου φαίνεται σαν να κρούμε το κόδωνα του κινδύνου και ας αναλογιστούμε πού ήμασταν. Αυτοματισμοί. Ένας αυτοματισμός που μπορεί να είναι υπολογίσιμος χωρίς να επιλύσει αποτελεσματικά μία κρίση, θα οδηγήσει σε προβλήματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι αυτοματισμοί αυτοί για να επηρεάσουν την αγορά. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι αν δεν προσέξουμε θα επιτύχουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Δεν πρέπει να είναι όργανο διαχείρισης κρίσης, αλλά Ε, ούτε να είναι μια σκούπα, ηλεκτρική σκούπα για χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε τι θα γίνει με την χρηματοδότηση, με την επαναχρηματοδότηση. Έχουμε εδώ αυτή την πρόταση. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο έχουμε όλο ένα και λιγότερα μέσα. Πώς θα το κάνουμε, ε, με, με ποιους πυλώνες, με τον πρώτο, με τον δεύτερο, από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα χρήματα. Τι επιπτώσεις θα έχουν εάν ελαττωθούν να επιστήσω την προσοχή σας. Δεν μπορούμε να ε, υπάρχουν κίνδυνοι εάν εμπλέξουμε πολλά μέσα-μέσα να δυσχεραθεί η κατάστασή μας. Επίσης, θεωρώ εξίσου σημαντικό ε, και σε, εξίσου κρίσιμο η, τον κίνδυνο να ενδυναμωθούν πάρα πολύ οι παραγωγοί. Πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργηθούν νέες ανισορροπίες ανάμεσα στους παραγωγούς και στους εμπόρους, ανάμεσα στους, ε, στις οργανώσεις των παραγωγών, τις ίδιες. Ήδη υπάρχουν εδώ κάποιες αντιρρήσεις. Επίσης, να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά νομικά συστήματα σε κάθε κράτος μέλος. Στη Γερμανία υπάρχουν, υπάρχουν, έχει διαφορετική αντιμετώπιση, υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί παραγωγών. Εάν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα όργανο διαχείρισης της κρίσης και δώσουμε χρήματα στην παραγωγή ή για παράδειγμα να δοθούν προϊόντα γάλακτος εκείνους που έχουν ανάγκη. Πρέπει να δούμε από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Έχω ακούσει πολλά ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό, να υποστηρίξουμε εκείνο, να ενισχύσουμε τον τάδε τομέα για μένα. Είναι επικίνδυνο για τον ε, προϋπολογισμό της Γεωργίας εδώ σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και τη διάθεση πόρων για τόσα πολλά πράγματα. Μετά, όσον αφορά για τον ε, κανονισμό και την επιμήκυνση των ποσοστώσεων της ζάχαρης ε, μέχρι το 2020, εδώ προτείνω να ακολουθήσουμε την Κομισιόν. Ο κανονισμός δεν έχει δεν είχε καλά αποτελέσματα ούτε στην αρχική ούτε στη διορθωμένη μορφή του. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να προσέξουμε να τον διορθώσουμε πραγματικά. Έπειτα χρειαζόμαστε τιμές αναφοράς ως μπούσουλα. Αλλά οι τιμές αυτές αναφοράς πρέπει να έχουν εξεταστεί και να έχουν εγκριθεί προσεκτικά και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι συνιστά αυτές τις τιμές, να συνεργαστούμε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο μαζί, Όμως η θέσπιση των τιμών είναι κάτι καθαρά τεχνικό, καθαρά μαθηματικό και αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει από την Κομισιόν. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η κρίση στην αγορά. Μιλάμε για κρίση. Αλλά πώς θα την ορίσουμε δικό μας, δική μας αρμοδιότητα είναι αυτή. Πρέπει να θέσουμε κριτήρια ορισμού μιας κρίσης. Η αντίδραση στην κρίση, το πώς θα γίνει αυτή η αντίδραση, είναι κάτι που είναι ήδη ρυθμισμένο στις ε, νομοθετικές πράξεις. Πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτές πραγματικά. Διότι εάν θέλουμε και αν θελήσουμε εμεί να ρυθμίσουμε τα πάντα, τότε θα έχουμε τεράστιο φόρτο εργασία. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Εν ολίγη αυτά είχα να πω. Θα ήθελα να ακούσω και του υπόλοιπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Συνάδελφοι, πάνω από 20 έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν. Λοιπόν, ε, σίγουρα η έκθεση Νταντέν είναι μια πολύπλοκη πρόταση. Έχουμε 400 τροπολογίες, αλλά δεν μπορούμε εμείς να τις συζητήσουμε μία προς μία θα πρέπει ο καθένας να μπει κατευθείαν στο ψαχνό όπου μπορούν να απαντήσουν και ο εισηγητής και η Κομισιόν. Ο Αντιπρόεδρος Μποβέ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά όταν έρχονται στην ώρα του στα τρένα δεν το συζητάμε καν, ενώ όταν αργούν γίνεται πάντα θέμα να ευχαριστήσω κατά πρώτον τον Μισελ για τη δουλειά του. Να πω ότι επέτρεψε τη συμμετοχή όλων των σχεδόν ε, εισηγητών στην επεξεργασία του κειμένου. Μας ενημέρωνε καθημερινά για το πώς εξελίσσεται το κείμενο και έτσι μπορέσαμε όλοι να ιδιοποιηθούμε τη σύνταξη του κειμένου. Οπότε να απηχηθούν και οι απόψει μα στο κείμενο που αναφέρεται στην ενιακό και να θεωρούμε ότι πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ήταν πολύ θετική αυτή η τάση. Δεν θέλω τώρα να σταθώ στα θετικά σημεία τη έκθεση, ακόμα και αν αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι έγινε πολλή δουλειά για τι ενώσει παραγωγών, για τι διαπαγγελματικέ ενώσει, με το άρθρο 106, 106α, 108. Εκεί υπάρχει πραγματικά μια δυναμική τάση που οδεύει στη σωστή κατεύθυνση από τα άρθρα 140 και 153 και για τις εξαιρέσεις των ε, ανταγωνιστικών δικαιωμάτων νομίζω ότι πραγματικά βρεθήκαμε εκεί στη δουλειά στην καρδιά της όλης δουλειάς, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα προβάλλει φραγμούς ε, στις διαπραγματεύσεις και γιατί δεν λειτουργούν σωστά η ΚΟΑ. Τώρα μπορούμε να θέσουμε στο επίκεντρο των ενδιαφέροντός μας την ανταγωνιστικότητα και τα δικαιώματα ανταγωνιστικότητα. οπότε ελπίζω ότι η Επιτροπή τη Γεωργίας θα ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, ότι θα μα ακολουθήσει και το Κοινοβούλιο και θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, όλα αυτά να ξεκινήσουν από την αρχή. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Επίση, για το θέμα της ε, αναταραχή τη αγορέ. εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ώστε να έχουμε εργαλεία που επιτρέπουν να δημιουργηθούν τέτοιε συνθήκε ώστε να διαχειριζόμαστε άμεσα τι κρίσει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας αποσχολήσει και πρέπει εκ των προτέρων να σκεφτούμε πού θέλουμε να καταλήξουμε. Αυτό δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη. Με το Ταμείο Αντασφάλισης και την ασφάλιση των εισοδημάτων. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει στο δεύτερο πυλώνα. Αυτή η συζήτηση είναι που πρέπει να γίνει με την αφορμή της έκθεσης Καπούλα Σάντο και εδώ είναι επί τη ουσία συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να αποφασίσουμε με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφισημία. Τελευταία ίσως, ε, τελευταίο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ, το ζήτημα των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς, διότι το πιο πρόσφατο παράδειγμα από την Γαλλία, με την κρίση των παραγωγών κρέατος πουλερικών, είδαμε ότι σήμερα αναταράξεις μπορεί να υπάρχουν ακόμα και τεχνητές. Εκείνοι το 65% των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων το χρησιμοποιούν για τα πουλερικά σε επίπεδο Γαλλίας. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Μία επιχείρηση σε 10 χρόνια έχει πάρει ένα θης ευρώ για να εξάγει προς τέτοιες χώρες. Νομίζω αυτό το είδος οι διαδικασίες πρέπει να πάυσουν. Διότι στις άμεσες εξαγωγές ερχόμαστε και προσθέτουμε και επιδοτήσεις για τα δημητριακά των ε, πουλερικών αυτών ακριβώ. Οπότε το σύστημα όπω δημιουργείται καταλήγει να είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη το τι ανάγκε έχει η αγορά, εφόσον θέλουμε να είναι απελευθερωμένοι, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν αυτέ τι πρακτικέ. Σε ευχαριστώ, Ζωζέ. Ο κύριο Κότα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Νταντέ για το εξαιρετικό του έργο. Τα ζητήματα αυτά και εμένα με απασχολούν ιδιαίτερα και συμμερίζομαι ιδιαίτερα στα δικαιώματα φύτευση, την παράταση ως το 2030, την εκχώρηση των δικαιωμάτων φύτευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν και οι νέοι που θέλουμε να ασχοληθούν με τη γεωργία να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους. οι, οργανώσει των παραγωγών, τρεις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, τις οποίες συμμερίζομαι. Απλώς να προσθέσω μια λεπτομέρεια. Σε πολλές από τις περιπτώσεις παραγωγής τροφίμων υπάρχει ανάγκη εποχιακής εργασίας. Στην Ιταλία υπάρχει μάλιστα το σύστημα των βάουτσερ για την πληρωμή αυτή της εποχικής εργασίας. Το 2009 ίσχυε σε, σε ένα μεγάλο βαθμό για τον πολιτικό τομέα και τον τρίγο και μετά επεκτάθηκε σε πολλούς κλάδους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να περιορίσουμε από τη μια την ε, παράνομη εργασία, αλλά να εξασφαλίσουμε και την απασχόληση κάποιων ε, εργαζομένων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Πολλέ είναι οι μονάδε που απασχολούν εποχικού εργαζομένου, όπω τα οποροκευτικά και τα αμπελουργικά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ποιε περίοδοι του έτου μα αφορούν και θα μπορούσαμε να πρέσουμε την πρόταση του συναδέλφου για τα οποροκευτικά και τα αμπελουργικά, ε, τον τομέα των αμπελουργικών, να προβλεφθούν αυτά τα βάουτσερ, ώστε να στηρίξουμε του εργαζομένου του τομέα. Ευχαριστούμε κύριο Ρούμπιξ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα αυτή την έκθεση που ήταν εξαιρετικά δομημένη και οργανωμένη σε κεφάλαια. Μας έδωσε μία πλήρη εικόνα των κυρίων προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με πολύ χαρά άκουσα ότι ε, αντιμετωπίστηκαν με σωστό τρόπο τα περισσότερα ζητήματα. Ωστόσο, η έκθεση προβλέπει οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε γεωργικά προϊόντα θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 20% και πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να συζητήσει την ε, πολιτική εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με την ΚΑΠ και το μέλλον της ΚΑΠ, διότι η αύξηση των εισαγωγών οπωσδήποτε θα επηρεάσει την ε, κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς. Δεν μπορώ να πω ότι, έχει, ότι έχουν εξισωθεί αυτές οι άμεσες ενισχύσεις σε όλες τις χώρες, διότι έχουμε τα νέα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στη Λετωνία, όπου οι γεωργοί αντιπροσωπεύονται κατά 50% λιγότερο σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Και οι άμεσες ενισχύσεις, για παράδειγμα στους ε, παραγωγούς λαχανικών, φτάνουν μετά από μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία και επίσης θα, πιστεύω θα έπρεπε να συζητήσουμε το ζήτημα των ποσοστώσεων της ζάχαρης. Εάν θέλουμε να τις κρατήσουμε μέχρι το 2020 ή ακόμα και το 2030, είναι κάτι που θα μπορούσα να το δεχτώ. Όμως η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα πιστεύει ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Τελείωσαν οι σκιώδεις εισηγητές, οπότε οι υπόλοιποι τρία λεπτά ο καθένας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τον οριζόντιο κανονισμό. Κανιέται και μετά άγνιο. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θαυμάζω την εξαιρετική δουλειά σας που βασίστηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή να ενισχυθεί η δύναμη των γεωργών στην αγορά. Επίσης, υποστηρίζω τις τροπολογίες για την ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών παραγωγών με τις διαπραγματεύσεις των τιμών, με τις συμβάσεις, με διαμεσολαβητικούς οργανισμούς. Διότι η γεωργία πρέπει να αποτελέσει μια εξαίρεση στον, ε, στους νόμους του ανταγωνισμού. έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των διαφορών σταδίων της γεωργικής παραγωγής. Ωστόσο, για τη ζάχαρη δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι το σύστημα των ποσοστώσεων θα έπρεπε να, επε... να επιμηκυνθεί μέχρι το 2020. Στην Λετωνία, εμείς θεωρούμε ότι το 2016 είναι μια κατάλληλη χρονιά να καταργηθούν οι ποσοστώσεις ζάχαρης, διότι θα ενίσχυε την παραγωγή ζάχαρης, θα μείωνε τις τιμές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εναρμόνιζε ε, περισσότερο τον τομέα της ζάχαρης με τις παγκόσμιες αγορές. Επίσης, ας σημειωθεί ότι 24 από τα 27 κράτη-μέλη αναφέρουν ότι υπήρχαν προβλήματα με την παροχή ε, ζάχαρης τα τελευταία χρόνια. Και μετά το 2015 δεν είναι απαραίτητο η ζάχαρη να είναι το μοναδικό αγαθό που θα εμπορεύεται με ποσοστώσεις. Έχει παρέλθει μια εποχή αναδιάρθρωσης από την τελευταία μεταρρύθμιση το 2006. Σε αυτό ε, στέκομαι, τα υπόλοιπα θα τα προτείνω ως δικές μου τροπολογίες στην έκθεση. Και ξανά να ευχαριστήσω τον κύριο Νταντέν για την εξαιρετική του δουλειά. E Ευχαριστούμε, Σάντρα. Κύριος Πρέπει να συγχαρώ τον Στίβεν Λαφόλ για την νέα του θέση στο Υπουργείο Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι είναι Γάλλος και σοσιαλιστής, εγώ τα πάω καλά μαζί του. Και θα συμφωνήσετε, πιστεύω κι εσείς, ότι είναι ο ομορφότερος άντρας αυτής εδώ της Επιτροπής προς απογοήτευση των ε, θηλυκών εδώ και των υπόλοιπων ψηφοφόρων. Τώρα, ο κύριος Νταντέν σίγουρα ε, συμπεριέλαβε την ζάχαρη στην έκθεσή του, όμως υπάρχουν πολλά σημεία που εξαφανίστηκαν. Για παράδειγμα, εξαφανίστηκαν 800, με αυτή την έκθεση 600 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βρετανική βιομηχανία επεξεργασία ζάχαρη δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Έτσι λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά βρίσκεται σε μία άσχημη θέση απώλεια κέρδου. Τα ζαχαρότευτλα και τα ζαχαροκάλα μας συνυπήρχαν για πάρα πολύ καιρό και ε, βοηθούσαν στην ευημερία των ε, αγροτών μας. Δυστυχώς η Κομισιόν έχει την δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση αυτή. Όμως, εάν θέλει να αλλάξει τις εξουσίες πρέπει να ελέγξει αυτούς που τις ασκούν. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος με την θέση της Βρετανικής κυβέρνησης για... και να διαφωνήσω με την απαλήφη των ποσοστώσεων, διότι αυτό θα ήταν κάτι καταστροφικό για τον Βρετανικό τομέα επεξεργασία ζάχαρης. Η Ελίζα και μετά Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά ευχαριστώ πολύ για τον εισηγητή, τον κύριο Νταντέν, γιατί πραγματικά παρουσίασε μια περιεκτικότατη έκθεση με πάρα πολλά επιμέρους σημεία, τα οποία θα μας προσανατολίσουν στο μέλλον της γεωργικής πολιτικής. Σίγουρα αναγνωρίζουμε όλοι ότι η γεωργία είναι σημαντικός τομέας της εσωτερικής ε, αγοράς και πρέπει να προσαρμοστεί στην ανταγωνιστικότητα. Ως εκ τούτου οι κανόνες επίσης πρέπει να, να εφαρμοστούν και στον τομέα αυτό. Πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος, είμαι πεπισμένη ότι είναι μια καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε, μπορούμε να εργαστούμε. Αλλά το ερώτημα είναι όπως ε, ε, διατυπώθηκε και πριν, για τις τιμές αναφορές. Ποια θα είναι η βάση των τιμών αναφοράς. Ποιο θα είναι το καθοριστικό σημείο για τον ορισμό των τιμών. Αναφέρθηκε ήδη το παράδειγμα. Αναφέρθηκαν οι δυνατότητες ε, αλλαγής των τιμών αυτών. Επίσης, η ενίσχυση των οργανισμών παραγωγών την θεωρώ κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους οργανισμούς παραγωγούς, παραγωγών. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ, ο Ούρλιχ και μετά τα Ραμπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Νταντέν και τον κύριο Ράτσεν. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία που μπορούμε να δούμε από αυτή την ε, έκθεση και αξίζουν τους επένους μας. Όμως εγώ θα επικεντρωθώ τώρα στα σημεία τα οποία θεωρώ προβληματικά. Έχω την εντύπωση ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 80 σε ορισμένα σημεία για τους οργανισμούς παραγωγών. Για, τα, για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η διαπραγμάτευση με τους εμπόρους να είναι δίκαιη. Μετά πρέπει να εφαρμοστούν ρυθμίσεις εάν υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές στις τιμές, μεγάλες αυξομοιώσεις. Ε, έπειτα το ζήτημα των νέων αγροτών που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά. Τι θα γίνει με εκείνους. Ε, θα βρεθούν σε πολύ μειονεκτική θέση εάν εξακολουθήσει να ισχύει η υπάρχουσα κατάσταση. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, πιστεύω ότι, θα, ότι είναι ένα όργανο αντιμετώπισης κρίσης και μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω. Για παράδειγμα, η αύξηση στο βούτυρο από 30 σε 70 χιλιάδες τόνους ε, είναι κάτι που θεωρώ προβληματικό και πραγματικά θέλω να κάνω έκκληση, να προσέξουμε αυτό το σημείο. Πριν από πολλά χρόνια ε, ακούσαμε ότι θέλαμε να ελαφρύνουμε το φόρτο των ε, παραγωγών βουτύρου και τώρα δεν μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό και να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρκ Ταραμπέλα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ Νταντάν και να τον συγχαρώ. Πρόκειται για ένα θέμα πρωτής της σημασίας. Τώρα, μερικά πράγματα χωρίς να είμαι εξαντλητικός δίκτυο ασφαλείας πρόκειται για μία λογική που θα πρέπει να την αναπτύξουμε για τους παραγωγούς στο σύνολό της και θα πρέπει να προβλέψουμε ή τιμές αναφοράς και η δραστηριοποίηση της ενίσχυσης προς αποθήκευση όπως επίσης και η συμβατότητα με τις ε, <coughs> τιμές αγοράς κλπ να γίνουν με διαβούλευση με τους ε, γεωργούς το ίδιο και για το γάλα και το ε, γάλα σε σκόνη με τις 30.000 τόνους αυτό το μου άρεσε Τώρα, για την παρακολούθηση της αγοράς από, την, ε, από το δημόσιο, ε, εδώ το συζητάμε, θέλει να υπάρχει ένας, μια ιδιωτική αύξηση του ρόλου των ιδιωτών. Ε, εγώ θα ήθελα όμως να έχουμε μεγαλύτερη αντιδραστικότητα στις διαταράξεις της αγοράς. Επίσης, για το θέμα της συνένωσης ε, των παραγωγών θα πρέπει, ε, θεωρώ ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, για το δικαίωμα του ανταγωνισμού, άρθρο 42 από τη συνδίκη της Ρώμης που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε και θα πρέπει να το γενικοποιήσουμε. Το αφήσαμε ανοιχτό εξάλλου και ως προπτική και στην έκθεση για το γάλα για τη γαλακτοπαραγωγή εκτίμησα για, λόγω των ε, σημαντικών ανισορροπιών στην αγορά του γάλακτος. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα τρία λεπτά πρόεδρε, να είστε ήσυχος. Για τις ανισορροπίες της ε, αγοράς ε, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών η ενίσχυση στους παραγωγούς που θα μείωνε εθελοντικά την παραγωγή και θα ε, έθετε και τα, το, τα πρόστιμα για όσους ξεπερνούν την παραγωγή, θεωρώ ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τη ζάχαρη. Σημερίζομαι την άποψη να συνεχίσουμε τις ποσοστώσεις μέχρι το 2005 όπως επίσης και συνέχιση των διαβουλεύσεων στον τομέα της αγοράς της ζάχαρης με τις αντιμαχίες που έχουμε στην Ευρώπη θα μπορούσαμε με την ενσωμάτωση των ποσοστώσεων να έχουμε μια ισορροπία στην αγορά. Το βιώνουμε σήμερα το πρόβλημα. Για το κρασί συμφωνώ απόλυτα για το 2030, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Για τα δικαιώματα φύτευσης, ε, αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των κρασιών, διατήρηση ε, του περιβάλλοντος, διατήρηση των οικογενειακών ε, παραγωγών. Όλα αυτά πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσω και μία δεύτερη φορά φαντάζομαι, αλλά δεν έχω σε αυτή τη φάση ειδικέ κριτικές ε, προς τον εισηγητή. επαναλαμβάνω τα συγχαρητήρια για τον ε, δρόμο στον οποίο εργάστηκε. Ευχαριστώ. Ο Λένι και μετά η Μάριαν Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και να τονίσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλύτερη σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο εισηγητής έχει προβλέψει πολλές λύσεις εξαιρετικές, οι οποίες μπορούν να αποσαφινιστούν ακόμη περαιτέρω, όπως ο ορισμός των τιμών αναφοράς, αλλά και η στήριξη των ενώσεων παραγωγών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ακριβώς αυτό το κείμενο μας δείχνει ότι από την αγορά αυτό που θα πρέπει να πρετανεύει στι μέρημνέ μα είναι η γεωργή. Η τελευταία δεκαετία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του γεωργικού κλάδου με την διαρκή μείωση των τιμών. Οι γεωργοί έχουν βρεθεί σε κατάσταση και σε συνθήκες κρίσης. Οι λύσεις που ως τώρα έχουν υιοθετηθεί δεν είναι δυστυχώς οι κατάλληλες, ακόμα και στον τομέα της ζάχαρης, όπως και των ε, γαλακτοκομικών. Οι διακυμάνσεις των τιμών ε, οδηγούν στο να δαπανώνται πολύ χρήματα για τις πληρωμές του γάλακτος, χωρίς όμως αυτά να καλύπτουν τις ανάγκες των παραγωγών. Άρα δεν ήταν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν το έγγραφο αυτό να λάβει υπόψη όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι για τις ποσοστώσεις της ζάχαρης και την παράσταση ως το 2020 πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μπορεί να έχουμε επικρίνει τις ποσοστώσεις της ζάχαρης και τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα αυτό, όμως δημιουργούνται πολλά προβλήματα από την ύπαρξη αυτή τη ποσόστοση στην αγορά. Εάν σήμερα θέλουμε να διτηρήσουμε το σύστημα των ποσοστώσεων, ε, γιατί αυτό να ισχύσει μόνο για το 2020, θα έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Ίσως λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί οι ποσοστώσει ζάχαρη δεν χρειάζονται καν. Ευχαριστούμε η Μαρέιντ. Και μετά κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, τα συγχαρητήριά μου προς τον εισηγητή. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο και μακροσκελές πόνημα αυτό. Τέλος πάντων ορισμένα σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την τροπολογία 391, για την παροχή βοήθειας σε παραγωγούς που οικειοθελώς διακόπτουν την παραγωγή και την ποινικοποίηση αυτών που, την τιμωρία αυτών που την αυξάνουν. Δεν καταλαβαίνω το συλλογισμό εδώ. Μου φαίνεται προβληματικός, διότι δύσκολο είναι η παραγωγή γάλακτος με ένα κουμπί να αυξάνεται ή να μειώνεται. Ε, θα χρειαστεί λοιπόν εδώ περισσότερη σκέψη και ανάλυση πριν μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την τροπολογία. να μειωνεται θα χρειαστει λοιπον εδω περισσοτερη σκεψη και αναλυση πριν μπορεσουμε να στηριξουμε αυτη την τροπολογια δευτερη μου παρατήρηση αφορά Τη ενό Παραγωγών και τι διαπαγγελματικέ ενώσει. που είναι πολύ ισχυρέ σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά καθόλου σε άλλα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ενιαίο μέγεθο για όλου. Δεν είναι η ίδια λύση κατάλληλη για όλου και θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Περαιτέρω, τρίτη παρατήρηση για τι ποσοστώσεις τη Ζάχαρη. Και άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν τι ανησυχίε του για την παράταση του συστήματο των ποσοστώσεων. Εμεί δεν έχουμε μετά τι τελευταίε ε, παραγωγή ζάχαρης. Θα πρέπει λοιπόν ο συγκεκριτή να σκεφτεί κατά πόσον τα κράτη-μέλη που εγκατέλειψαν την παραγωγή ζάχαρη μπορούσαν να διευκολυνθούν με κάποια ποσόστοση εάν παραμείνουμε στο σύστημα ποσοστώσεων στο 2020. Το έχει σκεφτεί αυτό καθόλου. Τέταρτη παρατήρηση, το δίκαιο ανταγωνισμού. Νομίζω εδώ χρειάζεται να δούμε πώς θα εφαρμόζουμε ενιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δίκαιο του αγωνισμού σε όλο τον τομέα της Γεωργίας υπάρχει ενιαία αγορά και η εσωτερική αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά. Νομίζω ότι οι τροπολογίε σα προ αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ευπρόσδεκτε αν θεωρούσαμε ότι θα ήταν αποτελεσματικέ. Θα ήθελα αυτό το σημείο να το συζητήσουμε. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι το στοιχείο αυτό τη μεταρρύθμιση τη ε, κοινή αγροτική πολιτική είναι εξίσου σημαντικό με τι άμεσε πληρωμέ. Θα χρειαστεί λοιπόν την ίδια προσοχή με αυτό του θέματος των αμέσων πληρωμών. Μιλάμε για τις μα... Ε, δομές ε, της ε, αγοράς και το πώς θα τη στηρίξουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον εισηγητή και να, τις ιδέες του και τις ερωτήσεις μου, το ίδιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κυρία Λούλιν και μετά κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ Νταντά για αυτή την τεράστια εργασία που αποτελεί μια σωστή βάση συζήτησης. Τρεις ε, σύντομες ερωτήσεις. <coughs> Μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Μαγκίνες σχετικά με την, με την πρόταση για το γαλακτοκομικό τομέα. Γιατί αναρωτιέμαι αν εδώ η πρόταση αυτή για να, έχουμε, να, να επανεισάγουμε την εισφορά δεν μου φαίνεται δηλαδή και πολύ εύκολο κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι από πού θα βρίσκαμε και τα λεφτά για τέτοιου είδους ε, επεμβάσεις. Ο κύριος Νταντέν μιλάει και για τη θνησιμότητα των μελισσών. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα για να έχουμε και την σωστή επιτυχία. Όλοι ζητάμε να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες των μελισσών μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκτινιατρικής πολιτικής. Για το δικαίωμα φύτευσης ε, των αμπελιών ξέρετε ότι θέλουμε να το διατηρήσουμε. Εγώ δεν θα άβαζα όμως ημερομηνίε. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το 2030. Θα έπρεπε απλώς ε, να ε, προασπίσουμε την διατήρηση του δικαιώματος φύτευσης και όπως επίσης και μία ευελιξία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Τρεις μικροπαρατηρήσεις λοιπόν είχα να κάνω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ, ο Χέρμπερτ και μετά ο Μάρτιν Χάουσλινγκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς τα βόδη. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια αναφερθήκαμε στις ποσοστώσεις του γάλακτος και πιστεύω ότι αυτό που μας πρότεινε η Κομισιόν τότε για τις ποσοστώσεις γάλακτος και για τα μέτρα αναδιάρθρωσης και για την προώθηση της εξόδου από αυτές τις ποσοστώσεις είναι αρκετά συνετά όμως δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν σε άλλους τομείς, για παράδειγμα τον, ε, την ε, γαλακτοκομικό τομέα στα, στις ορεινές περιοχές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ και ότι και πως αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και συμμερίζουμε την άποψη του συναδέλφου Νταντέν ότι πρέπει να αναλογιστούμε τι θα γίνει μετά από το 2015. Μετά το πακέτο για την ποιότητα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο τριμερούς διαλόγου και δεν, δεν προβλέπω να επιτύχει αυτός ο τριμερής διάλογος, καθώς φαίνεται. Είναι πολύ σημαντικό εμείς εδώ, στην έκθεση του κυρίου Νταντέν, να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να το επεξεργαστούμε στα πλαίσια του πακέτου για την ποιότητα, διότι δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο για αυτό το πακέτο. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Χέρμπερτ. Ο Μάρτιν. Και μετά ο κύριος Καπουλασάντος. Μάλιστα. Πραγματικά ο εισηγητή έκανε καλή δουλειά, μα έδωσε μπούσουλα σχετικά με το πώ πρέπει να πορευτούμε, από πού πρέπει να ε, αρχίσουμε και πραγματικά η άποψη για την ενίσχυση των ε, οργανισμών παραγωγών πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε ορισμένα ε, ζητήματα υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για μα, για παράδειγμα για την κρίση. Η κρίση Ελλάδα τα μπέρδεψαν, ναι, συνδέονται. Μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης λοιπόν. Την τελευταία εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε με την Επιτροπή και μας είπε ότι δεν υπάρχει κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Οι τιμές δεν είναι ακόμα σε στάδια παρέμβασης. Φυσικά πρέπει να έχουμε μηχανισμούς αντιμετώπισης της κρίσης, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται εγκαίρως. Και μας λείπει αυτό προς το παρόν. Μετά, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή για την ενίσχυση των παραγωγών και για έλεγχο των ενώσεων παραγωγών. Φυσικά είναι κάτι πολύ δύσκολο, πρέπει να οριστούν σαφείς κανόνες και ε, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν πολύ δυνατές αυτές οι ενώσεις παραγωγών. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πρέπει να δούμε τους ορισμούς, όπως αναφέρατε, για παράδειγμα, τους ορισμούς των συνεταιρισμών. Στην ε, Γερμανία το δίκαιο είναι διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες χώρες. Σε μια ένωση παραγωγών, η μια ένωση παραγωγών διαπέτει από άλλους κανόνες, όπως ε, αντί, σε σχέση με την Γαλλία, για παράδειγμα. Επίσης πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να επιμηκυνθούν οι διατάξεις για, το, για τον τομέα του κρασιού, για τα γαλακτοκομικά, για τα γαλακτοκομικά συμφωνώ και εγώ για, με όσοι υπόθηκαν για μετά το 2015. Όπως είπε και ο εισηγητής, το πακέτο για το γάλα δεν είναι αρκετό, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το 2015 Και δεν πρέπει να περιμένουμε τους, ε, τις ενώσεις παραγωγών, πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι μπορούμε να προσφέρουμε στους παραγωγούς, πώς θα αποζημιώνονται οι παραγωγοί που θα ε, παράγουν λιγότερα, λιγότερη ποσότητα. Πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα. Μετά, εξαγωγές, πρόθεση των εξαγωγών. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσαντες ότι χρειαζόμαστε ότι είναι ξεκάθαρο, ότι, ε, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ξεκάθαρη πολιτική εξαγωγών. Και με το να ψηφίσουμε θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Σε γενικές γραμμές Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για την μελλοντική συνεργασία με την Κομισιόν και ελπίζω σε καλό αποτέλεσμα. Λουίς, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους που συνεχάρισαν τον κύριο Νταντέν για το εξαιρετικό του έργο. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή βάση για να μπορέσει να βρεθεί μπαστική λύση με ευρία συνενέση από όλο το Κοινοβούλιο και χωρίς να πληγούν οι απόψει και τοποθετήσει των βουλευτών, συναδέλφων και των πολιτικών ομάδων. Θέλω λοιπόν να προσυπογράψω στι απόψει που εξέφρασε προηγουμένω η σκέδωση η συγκεκριά μα η Ράτσε. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω, το έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι, έχει να κάνει με τα γαλακτοκομικά. Όποιο βρέθηκε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα θα άκουσε ότι όλε οι παρεμβάσει, με ελάχιστε εξαιρέσει, Ίσως η κυρία Μαγκίνες να ήταν μία από τις λίγες φωνές κατά, μάλλον υπέρ της απελευθέρωσης του τομέα όπως προβλέπετε. Τέλος πάντων όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις ε, εξέφρασαν ε, σοβαρούς ενδιασμούς σε σχέση με τις επιπτώσεις της μελλοντική ε, απορρίθμισης της αγοράς. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να μας το παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο ο κ. Νταντά, αλλά είναι δύσκολο για λόγου δημοσιονομικού να υλοποιηθούν τα μέτρα που προτείνονται, όπω είπε ο συνάδελφο Λούλιν. Και υπάρχει και άλλο ζήτημα. Πώ θα στηρίζονται οι παραγωγοί που ε, προσωρινά αναστέλουν την παραγωγή του, δηλαδή οι παραγωγοί που κατά ένα χρονικό, ε, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πετάνε στα σκουπίδια τα, την παραγωγή του. Καθώ μια γελάδα δεν είναι κάτι που μπορεί να το προγραμματίσει κανεί με υπολογιστή για να βγάζει γάλα να μην βγάζει ή να σταματά να παράγει. Άρα Καταλαβαίνω ότι η θέση σας είναι κάπως ε, επιφυλακτική σε σχέση με τόσα προτείνονται με τα γαλακτοκομικά και τη ζάχαρη, όμως ε, λογικότερο θα ήταν να προτείνετε μέτρα ανάλογα με τον ίνο και τη ζάχαρη για το γάλα. Ε, καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να είστε κάπως μετροπαθείς εδώ, όμως λογικό θα ήταν εδώ να ακολουθήσουμε την εκπεφρασμένη θέση του Κοινοβουλίου, ώστε να είμαστε και πάλι προσεκτικοί σε σχέση με τη διακύμανση των τιμών, την αβεβαιότητα του μέλλοντος, ένα τομέα με τόσο μεγάλη σημασία και κοινωνική. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πιο προσεκτικά τον τρόπο που θα μπορούσαμε να ελέγχουμε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Ευχαριστούμε, Λουίς. Wow. Excellent timing. <laughs> Εξαιρετικός ε, συγχρονισμός. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νταντά για την ε, εισαγωγή του σε αυτήν την τόσο μακροσκελή έκθεση. Και θα ήθελα να λάβω αφορμή από τα σχόλιά του για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Είπε σε ένα σημείο ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο δικαίου ανταγωνισμού ερμηνεύεται διαφορετικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ήθελε λοιπόν προτάσεις από πλευρά μα για το πώς θα μπορούσαμε να, επεξεργαστούμε τέλος πάντων να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω. Στις κάτω χώρες υπάρχει το εξή ζήτημα. Συμφωνίες εντός τομέα, ενδοκλαδικέ ε, για την ευζοία των ζώων, τη βιώσιμη παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι γεωργείται περισσότερα στην ίδια του την εκμετάλλευση. Γιατί με τα εργοστάσια, τι αγορέ, του εμπροδομένου, έχουν ε, συμφωνήσει να βελτιώσουν ε, τα πρότυπα ευζοία των ζώων ή τα περιβαλλοντικά και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή όμως οι γεωργοί έχουν επιστροφή των επενδύσεων μόνο με υψηλέ, υψηλότερες τιμές, αύξηση των τιμών και όχι με αύξηση του περιθώριου κέρδους τους. Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγεί σε συμφωνίες που να συμπεριέχουν και την ε, συνιστόσα τη τιμή. Πράγμα που δεν γίνεται αυτή την ώρα. Δεν καλύπτω το ολόκληρη αλυσίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Θα ήθελα λοιπόν να επεξεργαστούμε με τον κύριο Νταντά λύσει για το πώ μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι αυτού είδου οι συμφωνίε που να καλύπτουν όλη την αλυσίδα παραγωγή από την εκμετάλλευση ω το πιάτο του καταναλωτή όχι μόνο επιτρέπουν και την, τα ποιοτικότερα προϊόντα, αλλά και καλύτερο περιθώριο για του γεωργού. Διότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται αυτέ οι επενδύσει, εάν στο τέλο το περιθώριο των ε, γεωργών δεν ε, βελτιώνονται. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή τα περιθώρια ποια είναι στου περισσότερου τομεί τη γεωργία. Θα συνεργαστώ λοιπόν μαζί του για να του πω τι ιδέε μου, ευχαρίστω. Και ο κ. Νταντά ζήτησε τι συνεισφορέ μα. Άρα από μένα θα τι έχει. Και να ολοκληρώσω λέγοντα ότι νομίζω η μέγιστη πρόκληση εδώ κατά τη συζήτηση τη αγροτική πολιτική, είναι να βεβαιωθούμε ότι έχουν καλύτερε τιμέ οι γεωργοί. συζητούμε κατά λεπτό πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τη μεταρρύθμιση τη αγροτική πολιτική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δούμε και το θέμα τη πολιτική ανταγωνισμού. Ίσως είναι και σημαντικότερο διότι όταν ή εάν η γεωργία απελευθερωθεί περαιτέρω, εάν οι τιμέ ή μάλλον τα κονδύλια διαρκώ μικραίνουν για την ΚΑΠ, πράγμα που ήδη συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τον ανταγωνισμό και τι τιμέ πολύ περισσότερο. Ανυπομονώ λοιπόν να ε, συνεργαστούμε τον κύριο Ταντά για τα θέματα αυτά και έχω και μια ερώτηση για τη ζάχαρη. Προτείνει την παράταση του συστήματο προσωστώσεων στο 2020. Δεν είμαι και θειαζότρια των ε, ποσοστώσεων, αλλά μπορώ να τον στηρίξω σε αυτό και καταλαβαίνω ότι στο ενδιάμεσο θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη πρόοδο. Όμω, με τι εκθέσει τι θα γίνει στο 2018, διότι φοβάμαι κάπω ότι αν έχουμε εκθέσει που θα με τις οποίες θα διακυβεύεται το αν θα συνεχιστεί ή όχι το σύστημα των ποσοστώσεων, θα είναι δύσκολο να θέσουμε τέρμα κάποια στιγμή. Άρα επεξεργαζόμαστε το τι θα γίνει με τις γαλακτοκομικές ε, ποσοστώσεις από το 2014 είναι η τελευταία προθεσμία. Ξέρουμε πώς θα γίνει η μετάβαση στο νέο σύστημα. Ε, είμαστε προετοιμασμένοι. Ή το 2018 θα έχουμε μια έκθεση για να αποφασίσουμε τελικώ εάν το σύστημα θα αλλάξει ή όχι. Διότι σε αυτή την περίπτωση μέχρι το 2018 μπορούμε να αποφασίσουμε να μην αλλάξει και ποτέ. Ευχαριστώ, George Leiden. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον Μισελ Ταντέν για την λεπτομερέστατη και ογκοδέστατη έκθεση και τις τροπολογίες του. Καταρχάς, καλωσορίζω την σοβαρή του προσπάθεια να πολεμήσει το Συμβούλιο και την Κομισιόν στο, στην προσπάθειά τους να πάρουν εξουσίες από το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιώντας πράξεις, ε, εφαρμοστικές πράξεις αντί για πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν πρέπει να είμαστε σαφείς στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τις εξουσίες μας. Όσον αφορά την παρουσίαση του Μισελ Τόλα διακρίνω μία αναφορά, στις, ε, μία επιστροφή στις ημέρες της ε, έντονα ρυθμιζόμενης αγοράς, οι οποίες είχαν μεγάλη ωφέλη για τους παραγωγούς και αναρωτιέμαι και αν ε, αυτές οι προτάσεις ενισχύουν πολύ, περισσότερο από όσο θα έπρεπε τους παραγωγούς. Εμείς ως Κοινοβούλιο οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την θέση των παραγωγών στην αγορά, ώστε να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή τιμή για τα προϊόντα τους, χωρίς όμως να ξεπεράσουμε τα όρια, χωρίς όμως να τιμωρούμε τους παραγωγούς που παράγουν ε, μεγαλύτερες ποσότητες Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στις, ε, στην επιχείρησή τους, έχουν γίνει πιο αποδοτικοί, έχουν επεκταθεί. Δεν θα πρέπει αυτή να εμποδίζονται, να εμποδίζεται η επιτυχία τους. Βασισμένοι λοιπόν σε αυτό, θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά τις προτάσεις του Μισελ και θα ε, προσπαθήσουμε να αποφανθούμε για το αν ενδυναμώνει την θέση των παραγωγών στην αγορά ή εάν παρεμβαίνει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νταντέν στο τέλος εάν έχει χρόνο, να, ε, εάν μπορεί να μας ε, αποσαφηνίσει το άρθρο 106, την τροπολογία 106 και πώς θέλει να επιφέρει μία ισορροπία, δηλαδή στους παραγωγούς που θα ανταμείβονται, τι θα γίνει με τους παραγωγούς που βρίσκονται πάνω από τις ποσοστώσεις, με αυτούς που βρίσκονται κάτω από τις ποσοστώσεις θα υπάρχει ποινή για όσους επερβαίνουν τις ποσοστώσεις, ανταμοιβέ. Επίσης τι θα γίνει με τις ποσοστώσεις του γάλακτος. Γιατί πιστεύω ότι οι απόψεις σας για τις ποσοστώσεις γάλακτος είναι αρκετά ενδιαφέροντες. Ευχαριστώ. Εδώ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και ήθελα να το τονίσω αυτό. Να πω ότι λόγω χάρη η ενίσχυση των ενώσεων παραγωγών είναι ουσιαστική σημασία και πρέπει να γίνει όχι μόνο για την ενώσεις ενώσει παραγωγών, αλλά οπωσδήποτε και για αυτέ που ήδη υπάρχουν. Αυτό μου φαίνεται μια πτυχή καθοριστική. Να τονίσω και το εξή. Αυτό που χρειαζόμαστε στην ε, ενιαία ΚΟΑ και για τους γεωργούς και για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας είναι να προχωρήσουμε στην σταθεροποίηση των αγορών και σε μια εξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων που ήδη υπάρχουν στις αγορές αυτές με τις νέες γεωργικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Εδώ επικεντρώνεται και ο ρόλος της ενιαίας ΚΟΑ. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το εξή. Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μόνο τα μέσα που προβλέπονται, αλλά και για το μέλλον, αλλά να προβλέψουμε και ρυθμιτικές διατάξεις αναδρομικά. Δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή του γαλακτοπαραγωγικού τομέα, δεν υπάρχει εκεί ισορροπία προσφοράς ζήτησης οπωσδήποτε. Κάποια αφορά λοιπόν η ύπαρξη προϊόντων, η διάθεση προϊόντων οδηγεί στην εξαγωγή τους με πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό πλήττει τους παραγωγούς. Αυτό είναι το σημερινό σκηνικό. Πίεση στο κόστος και διακύμανση των τιμών. Δεν, ε, οι πρώτες ύλες δεν λείπουν τα τρόφιμα ή τα ζώα. Όμως η πτώση των τιμών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εξακολούθηση της λειτουργίας κάποιων εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την παραγωγή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι εμπορικές παρεμβάσεις και η διανομή. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με το θέμα της δικαιοσύνης, πολύ περισσότερο σημαντικό είναι αυτό, διότι αν για παράδειγμα στην Πορτογαλία πραγματικές τιμές έχουν μειωθεί κατά 26% από ότι, περισσότερο από ό,τι συμβαίνει, αυτό ε, σημαίνει ότι μπορεί το κόστος να είναι χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, άρα οι γεωργοί δεν καταφέρουν να φτάσουν στην αγορά και να καλύψουν το κόστος τους. Οπότε, αν δεν περάσουν από την αγορά, η έλλειψη ισορροπίας οδηγεί στο τα σημερινά περιθώρια να είναι πολύ σφιχτά, ώστε να ε, ε, αντισταθούν στην πτώση των τιμών. Άρα, είναι καθοριστική σημασία να το σκεφτούμε αυτό για την επιβίωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Και κάτι άλλο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό είναι να δούμε το θέμα των εμπορικών συμφωνιών. Διότι η γεωργία δεν μπορεί να είναι ένα νόμισμα συναλλαγής και ισοτιμίας. Θα πρέπει να υπάρχει ε, εμπορική δικαιοσύνη και αυτό να επιτρέψει στην γεωργία μας να είναι και ανθεκτική ε, στο επίπεδο του ΠΟΕ. Ευχαριστώ Λουίς, Φαϊμό και μετά Γιάρ. Και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου για την επέκταση, για την επιμεκίνηση της ποσόστοσης ζάχαρης. Στην Τσεχία οι ποσοστώσεις αυτές δεν έχουν φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει και για την τελευταία μεταρρύθμιση. Η, αύξηση, η τιμή της ζαχαρής έχει αυξηθεί. Και αυτό δεν είναι καλό για τους παραγωγούς ζάχαρης. Έτσι λοιπόν διαφωνώ με την επιμήκυνση του καθεστώτος με την επιμήκυνση των ποσοστώσεων της ζάχαρης, διότι χωρίς αυτές τις ποσοστώσεις η αγορά πιστεύω πως θα λειτουργεί καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει το 2016. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή γιατί μας προτείνει να επιμηκυνθούν αυτές οι ποσοστώσεις και πέρα από τότε. Διότι το καθεστώς της ε, ζάχαρης σήμερα, έτσι όπως είναι, δεν βοηθά ούτε τους καταναλωτές, ούτε τους παραγωγούς, ούτε τις εταιρείες που ε, παραγωγής ζάχαρης, ε, ούτε αυτές έχουν κάποιο κέρδος. Γιατί λοιπόν να το συνεχίσουμε. Πέτρα Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο, γι' αυτό λοιπόν θα είμαι σύντομο με τις ευχαριστίες. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, για τις ε, ενώσει παραγωγών χρειάζεται ορισμός. Το πλαίσιο πρέπει να το ορίσουμε σαφέστατα. Δεν, δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά αυτό. Υπάρχουν πολλά επιμε, πολλές ιδιαιτερότητες σε κάθε κράτος μέλος. Και Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο και τότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν θα, είναι, θα παραδυναμώσουν αυτές οι ενώσεις παραγωγών. Μετά για τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς. Έχουμε δύο μέτρα επιρροής της αγοράς αυτή τη στιγμή. Δύο δυνατότητες, την αποθήκευση και τις επιδοτήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ε, ε, υποστηρίζω να, εφαρμόσουμε και τα δύο όργανα αυτά. Όμως η ερώτησή μου είναι από ποιο σημείο και μετά επεμβαίνουμε, από ποια τιμή και έπειτα. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ας προσέξουμε να μην γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80, στην αγροτική πολιτική της δεκαετίας του 80. Δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο μόνο εάν υπάρξουν σημαντικές ανισορροπίες στην αγορά θα έπρεπε να επέμβουμε. Διότι όντας πολύ παρεμβατικοί θα δώσουμε άσχημα, άσχημα σινιάλα στην αγορά. Έπειτα για τη ζάχαρη. Προβλέπετε κάτι για το βαμβάκι, για την αγορά βάμβακος. Θέλουμε να συνεχίσουμε με την αγορά φάρμακος έτσι όπως έχει, θέλουμε να την αλλάξουμε. Τι θα γίνει εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντές έχει το λόγο. Και για εκ μέρους της δικής μου κοινοβουλευτικής ομάδας θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Νταντέν για τις 300 σελίδες, 320 σελίδες της έκθεσής του. Έχουμε, έχω, έχω παρατηρήσει θετικές αλλαγές διαγράφηκαν 24 άρθρα, υπάρχ, ε, ξαναγράφτηκαν 107 τροπολογίες, όμως το έργο μας είναι να είμαστε επικοδομητικοί και να συμβιβαστούμε στις τροπολογίες, να προσπαθήσουμε με αυτές να βελτιώσουμε την νέα αγροτική πολιτική. Τώρα όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις και, την, και τις τεχνικές επιπτώσεις. Δεν είμαι σε θέση να επεκταθώ, πρέπει να το, να το εξετάσουμε. Όμως πιστεύω, όπως και η Μπρίτα Ράιμερς, ότι χρειαζόμαστε πολιτικές αποφάσεις και όχι αυτοματισμούς. Ελάχιστο παρεμβατισμό, αλλά σαφής, σαφές πλαίσιο, ενισχύσεις, όπου είναι αναγκαίο. Όταν ε, αναφέρατε πως 70.000 τόνοι για παράδειγμα είναι υπερβολική. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η ποσότητα αυτή θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν θέλουμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης. Δεν θα κοστίσει πολύ στους φορολογούμενους εάν αγοράσουμε σε πιο χαμηλές τιμές και μετά περιμένουμε να αυξηθούν και προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αυτές τις τιμές. Τώρα όσον αφορά τη ζάχαρη, και το κρασί. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση του κυρίου Νταντέν. Οι καταναλωτές πρέπει να πληρώνουν αυτή τη στιγμή ψηλότερες τιμές. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την τιμή της ζάχαρης. Διότι όπως είδαμε υπάρχουν πάρα πολλοί, αγρο... Ε, πολλοί παραγωγοί ζάχαρης που έχουν σταματήσει να παράγουν ζάχαρη. Διότι είναι πολύ ακριβή, διότι μπορούν να την, αγοράσουν, να την αγοράσουμε πολύ φτηνά από την Βραζιλία ή από την Κίνα, για παράδειγμα. Υποστηρίζω την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών επίσης. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση των παραγωγών. Στόχος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχουμε μηχανισμούς αντιμετώπισης της κρίσης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ευπορία των πολιτών μας. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Να συγχαρώ για τα εξικοστά του γενέθλια τον αγαπητό μας συνάδελφο και να πω στην Αυστρία στην Αυστρία η ποσότητα. Υπάρχουν διαφορές στην Αυστρία και στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά τις, τις ε, ποσότητες κατανάλωσης της, ε, ποσότητες κατανάλωσης βούτυρου που ενδείκνυται. E Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο, τον κύριο Νταντέα, για το διτάνιο έργο του. Έγιναν πολλές ορθές παρατηρήσεις επί των λεπτομεριών. Δεν θα ήθελα να παραμείνω σε αυτές. Έχω όμως μια γενική παρατηρήση. που βρίσκονται και σφαιρικό χαρακτήρα. Έχει και κανείς άλλος δεν την ανέφερε τώρα. Ως Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου θα κληθούμε να απαντήσουμε σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές ερωτήσεις για τον συνολικό προσανατολισμό αυτής της έκθεσης. Δεν λέω ότι εγώ διαφωνώ με τον προσανατολισμό αυτό, όμως δεν έχω καμία αντίρρηση για την προστασία τη Ευρωπαϊκή Γεωργία, ιδίω των γεωργών και των κοινοτρόφων. Αυτή είναι η δουλειά μα, άλλωστε. Αυτό που με ανησυχεί είναι, και αν καλά κατάλαβα την αισθέτη εδώ, νομίζω ότι επαναλαμβάνω και τι δικέ τη ανησυχίε, είναι εάν τελικά έχουμε ένα μικρότερο και πιο περιορισμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο τελικό αποτέλεσμα. Πώς στο καλό θα καταφέρουμε να βρούμε χρήματα για όλα αυτά, πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση δεν θα είναι τόσο ευχάριστα και ήρεμα τα πράγματα τότε. Ορίστε. Αυτό ήθελα να ακουστεί. <clears throat> Ευχαριστώ όλους σας. Εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Πατσέκο, στον Διευθυντή και μετά ο Μισελ Νταντάν για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νταντάν τον εισηγητή για μια έκθεση που είναι και πολύ αναλυτική αλλά και σε βάθος εξετάζει όλες τις πλευρές της ενιαίας ΚΟΑ και τις μεταρρυθμιστικές μας προτάσεις. Δεν θα σταθώ σε όλες τις τροπολογίες, δεν είναι ο κατάλληλος τόπος, ούτε έχω και το χρόνο. Θα ήθελα όμως να πω μερικές πρώτες αντιδράσεις για σημαντικά πράγματα. Για τις οργανώσεις των παραγωγών, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συμμεριστούμε απόλυτα τις επιθυμίες του εισηγητού του κυρίου Νταντά. Δηλαδή, να έχουμε μία ενίσχυση της θέσης των παραγωγών μέσα στο όλο δίκτυο, μέσα στον όλο κλάδο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε Τώρα πιστεύω ότι και ο ίδιος εξαλλού το αναγνώρισε, πρέπει να ενισχύσουμε το δίκτυο χωρίς όμως να δημιουργήσουμε ένα καρτέλ, μια καρτελοποίηση. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενίσχυσης των οργανώσεων των παραγωγών και των θεμάτων του δικαίου ανταγωνισμού σχετικά με τις ερωτήσεις για το δίκτυο ασφαλείας και την οργάνωση των αγορών. Εγώ σημειώνω ότι ο κύριος Νταντά διατηρεί επί της ουσίας τις ε, θέσεις ε, της ε, ΚΑΠ για τον προσανατολισμό της αγοράς. Προτείνει ορισμένες τακτοποίησεις θα έλεγα όμως ότι για αυτές τις τακτοποίησεις θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, να τις δούμε από κοντά. Υπάρχει όμως ένα σημείο πολύ σημαντικό για το οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Εμείς εκτιμούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τις κρίσεις των αγροτικών αγορών είναι τα εξαιρετικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα. Γιατί, Γιατί είναι ευέλικτα, προσαρμόζονται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των κρίσεων, χωρίς τεχνητά να δημιουργούμε διέξοδα της αγοράς ε, με αύξηση των τιμών αναφοράς. Έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και όχι μία πολιτική που στα τυφλά θα αύξανε τις τιμές αναφοράς. Πράγμα το οποίο εξάλλου δεν το προτείνει καν ο κύριος Δαντά. Ένα άλλο σημείο το οποίο διαπιστώσαμε, το οποίο θύχτηκε εδώ, Είναι ένα σημείο το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις μας. Ποσοστώσεις για τη ζάχαρη. Ο κύριος Νταντά επανισάγει τις ποσοστώσεις ε, ζάχαρη, για τη ζάχαρη στο σύστημα της ε, Νέας ΚΟΑ. Ήρθε η ώρα ο ζαχαροκομικός ε, κοτομέας να καρποθεί των ευκαιριών που δημιουργούνται με την αύξηση της ζήτηση στις διεθνείς αγορές. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κλειστεί σε ένα καλούπι και να μην ε, εκμεταλλευτεί τις ε, ε, ευκαιρίες που το δίνονται. Μέσω της διεθνούς συγκυρίας εμείς αυξάνουμε βάσει αυτών των συμφωνιών τις εισαγωγές μας και δεν επιτρέπουμε σε αυτόν τον τομέα να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια αγορά εμείς θεωρούμε ότι ε, ε, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα ο κλάδος. Θα μπορούσε λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αφορά στις προτάσεις μας αλλά θύχτηκε και συζητιέται Ο κύριος Τσόλος, ο Επίτροπος, σύστησε μία ομάδα υψηλού επίπεδου για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του βουλευτού ο οποίος ζητεί την παράταση των δικαιωμάτων φύτευσης χωρίς όμως να αλλάξουν οι κανόνες στον τομέα και χωρίς να αμφισβητηθούν και οι δυνατότητες επέκτασης του τομέα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά Πατσέκο θα έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία. Μίσελ, θέλεις να πεις μερικά τελικά. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις ευχαριστίες σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά, διότι οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν παρόμοια θέματα. Για τη ζάχαρη. Να είμαστε ειλικρινεί. Σε αυτό το σώμα βρισκόμαστε όλοι και συμμετέχουμε εδώ και τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της τριετίας από κοινού ψηφίσαμε κάποιες εκθέσεις, ιδίως την έκθεση Lion και DES, που ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία. Την έκθεση DES την ψηφίσαμε τον Ιούνιο 2010-2011 μάλλον. Εκεί υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένε θέσεις. Δεν μπορώ τώρα εγώ να ε, ε, υιοθετήσω αντίθετε θέσει με την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τη ζάχαρη ε, ψηφίσαμε πριν από ένα χρόνο, ζητώντα την παράταση ω το 2020 του συστήματο ποσοστώσεων. Είναι μια θέση ελλημένη. Ε, το 2020 ε, για την νέα θήτευση συμφωνώ με όλου του ε, με παρενέβησαν διότι παράλληλα με την αναθεώρηση του κειμένου θα ληφθούν απόψη τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου ιδίω στο σημείο αυτό του κειμένου, για το γάλα. Ίδιο ζήτημα και ίδια, ίδια περίπτωση. Ακριβώ πριν, κατά τη διάρκεια τη τριετία, το κοινοβούλιο τοποθετήθηκε κατά των ποσοστώσεων του γάλακτο. Τώρα δεν μπορούσα να αμφισβητήσω ή να προωθήσω ένα επιχείρημα που θεωρούσα ότι ήταν εξ αρχή ζητημένο. Εάν υπάρχει πλειοψηφία βεβαίω, ευχαρίστω στη νέα πλειοψηφία που θα έχει δημιουργηθεί να τη λάβω υπόψη. Μου φάνηκε πιο συνετό να υποβάλω μια πρόταση που κατά την άποψή μου να προκαλέσει συζήτηση. Θεωρώ ότι επιδέχεται βελτιώσεων. Είναι μια πρόταση που θα πρέπει να εξισορροπηθεί ώστε να γίνουν δαπάνε ω προ τι χρηματοδοτήσει. Με σκοπό όχι να πάυσουν οι παραγωγοί την παραγωγή του, αλλά να αντισταθμιστεί η παραγωγή του 10-15-20%. Να σα θυμίσω ότι έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία φορά. Όταν υπήρξε κρίση γάλακτο την περασμένη φορά, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί μείωσαν την παραγωγή και τα περιθώρια κέρδους αναζητήθηκαν από τους μεγάλους παραγωγούς και διανεμήθηκαν στους υπόλοιπου για να εξισορροπηθεί η κατάσταση στην αγορά. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα στα οποία κλήθηκα να απαντήσω. Δεν έχω να πω κάτι στην παρατήρηση ότι είναι ατελής η πρότασή μου, γι' αυτό και περιμένω τις τροπολογίε για να βελτιωθεί. Τώρα για το θέμα τη διαχείριση των αγορών, την παρέμβαση, την αποθεματοποίηση και το καθεξή. Άκουσα τι παρατηρήσει κάποιων από εσά και είπατε ότι φοβάστε μήπω αναστηθεί το παρελθόν. νομίζω ότι είμαστε όλοι στη δίμηκο Κοιτάξτε, α δούμε μελό μαζί. Πού βρίσκεται το δίκτυο ασφαλεία που προβλέπουμε. Ποιε είναι οι τιμέ αναφορά, ποιε είναι οι τιμέ παρέμβαση, 80% των τιμών, 90% μάλλον των τιμών αναφορά. κάτι που επιτρέπει παρέμβαση σε περίπτωση καταστροφής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολλοί παραγωγοί στην Ευρώπη που είναι ικανοί να έχουν εισόδημα ικανό με την τιμή παρέμβαση. Η τιμή παρέμβασης για το σύτολο που χάρη. Είναι 90 ευρώ τόνο. Η τιμή παρέμβασης για το κρέα είναι 2.000 ευρώ τόνο επειδή με παρέμβασε για το γάλα και θα μπορούσα να συνεχίσω έτσι να παριθμώ παραδείγματα. Στην πραγματικότητα όμω δεν είναι μηχανισμοί που σκοπό έχουν να αναδημιουργούν αποθέματα, αλλά την ε, διαχείριση κρίσεων θέλουν να εξασφαλίσουν ώστε να αποφύγουμε ενδεχόμενε καταστροφές. Νομίζω δεν θα ήταν και φιλοσοφικός ορθό αυτή τη στιγμή να να χρησιμοποιήσουμε ξανά εργαλείο του παρελθόντος. Για το Βάμπακα. Θα απαντήσω εν καιρό τώρα για τα απορροκυπευτικά στην σχέδιο συγκεκριά μας να πω ότι το άρθρο 89 ε, ε, ανταποκρίνεται και στο 88 που παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για τα απορροκυπευτικά και προσθέτει στην μπανάνα και τα επεξεργασμένα φρούτα. Είναι λοιπόν το επόμενο άρθρο που αναγκαστικά λαμβάνει υπόψη την προσθήκη του προηγούμενου. Για όσα πρότεινε ο Λορέντ, Ε, θα είναι ευπρόσδεκτε οι προτάσει και οι δικέ του και όλων των υπολείπων που στι ερχόμενε ώρε θα θελήσουν να αποβάλουν νέε τροπολογίε. Ε, ευχαριστούμε, Μισελ. Να θυμίσω στου συναδέλφου για την έκθεση του Μισελ. Η προθεσμία βολή τροπολογιών λήγει στι 10 Ιουλίου στι 12 το μεσημέρι. Θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά είναι ένα σημαντικό έργο που θα περάσει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα πρέπει να δούμε μάλιστα το τέλο τη τροπολογία. Έχουμε πραγματικά λοιπόν με τη δουλειά του Μισελ να μπορέσουμε να παραμείνουμε με λίγε και ξεκάθαρε τροπολογίε. Περνάμε στο σημείο 5. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση τη της ε, κοινή γεωργική πολιτική. Συγκητή ο κ. Λαβία η πρόταση του οριζόντιου, της μέτρων για τη μεταρρύθμιση είναι πάλι το θέμα μας και να θυμίσω εδώ ότι για τον κύριο Λαβία και την έκθεσή του η προθεσμία υποβολής τροπολογιών λήγει στις 9 Ιουλίου στις 12. Θα μείνει μαζί μας ο διευθυντής Πατσέκο. Τζοβάνι, στο λόγο για την παρουσίαση. <coughs> Ευχαριστώ Πρόεδρε, έτσι όπως έπραξες εσύ αλλά και ο συνάδελφος Νταντέν θα εξάρω κι εγώ τη σημασία της ημέρας ε, όπου το κοινοβούλιο παρουσιάζει τους καρπούς της εργασίας του. Εργασίας μέσα σε ένα νέο πλαίσιο μαζί με τον Νταντέν και τον Κάπουλα στους άλλους εισηγητές προτείνουμε τις απαραίτητες κλίδες για ή το άνοιγμα των νέων ευκαιριών των Ευρωπαίων γεωργών που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Πρέπει να βρούμε από κοινού τη διαδρομή που θα μας οδηγήσει σε μια συμμερισμένη ΚΑΠ που δεν θα αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των γεωργών μας. Σημερίζομαι ότι οι τέσσερις προτάσεις θα πρέπει να αποτελέσουν τα μέσα για να εφαρμόσουμε σήμερα τα αιτήματα εκείνα που προβάλλουν εδώ και πολύ χρόνια οι Γεωργοί. Και μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας υποχρέωσή μας είναι να τους ακούσουμε, να τους καταστήσουμε ενεργούς ε, στην όλη συζήτηση για να έχουμε μετρημένα αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο μέσα από την έκθεση πρωτοβουλίας του Άσφορτ για την απλούστευση της ΚΑΠ εκφράστηκε τον Μάιο του 2010 ως προς το κατεπήγον της ανάγκης του να γίνει πιο εύκολη η ζωή των Γιωργών. Αυτή την απέτηση την τονίσαμε πολλάκις με την έκθεση Λάιον του 2010 και του ΝΤΕΣ το 2011 όταν το Κοινοβούλιο επικύρωσε τη βούλησή του και τη στράτευσή του για να απλουστευτεί ο σύνθετος διοικητικός μηχανισμός και να μειωθούν οι δαπάνες εις βάρος των γεωργών και μετά την ΚΑΠ του 2013. Εγώ ξεκινάω από αυτήν την ανάγκη απλούστευσης της ΚΑΠ <coughs> για να σας αναφέρω ποιες είναι οι βασικές προτάσεις τροποποίησης στην πρόταση που διατυπώνει η Κομισιόν. Υποστηρίζω, όπως πάρα πολλές φορές είπαμε σε αυτήν την Επιτροπή, ότι απλούστευση σημαίνει μη κατασπατάληση του ελευθέρου χρόνου των Γιωργών. Θεωρώ απαραίτητο να προτείνω μία ουσιαστική αλλαγή σε αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν στην πρόταση κανονισμού, δηλαδή δυνατότητα οι γεωργοί να μπορούν να παρουσιάζουν για την ενιαία πληρωμή όπως και για τις άλλες αιτήσει τους ένα αίτημα με, με πολυετή διάρκεια και ετήσια επικύρωση, επιβεβαίωση. Δηλαδή όσοι δεν, δεν αλλάζουν την γεωργική τους επιχείρηση θα υποβάλουν μία αίτηση με πολιετή διάρκεια. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε και, να έχουμε και την προσφυγή στην τεχνολογία, έτσι όπως το προτείνει ο εκτελεστικός κανονισμός της Κομισιόν 365 του 12, για να αποφύγουμε η πολλή χαρτούρα να εγκλωβίζει, να παρακολεί τη δραστηριότητα του Γιώργου. Προς την ίδια κατεύθυνση τίνει και η πρόταση που διατυπώνω για την αλλαγή της τεχνικής βοήθειας προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για την Κομισιόν οι υπηρεσίες που προσέφεραν οι που προσέφερε τεχνική βοήθεια αφορούσε στην αιρεσιμότητα και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εγώ θεωρώ όμως ότι η γκάμα των προσφορών μπορεί να μεγαλώσει και αναφέρω εδώ και εκείνη την απαραίτητη υποδομή για να πάμε προς την αγορά. Εγώ με τις τροπολογίες μου προσπάθησα να καταστήσω διαφανές το θέμα των κυρώσεων προς τους γεωργούς που δεν είναι και πολύ ευχάριστο για τους γεωργούς, αλλά θα πρέπει να είναι κατανοητό από όλους για να αποφύγουμε οι γεωργοί να μην ε, ε, κάνουν παραβιάσεις. Αυτό αφορά και στην πρόταση συναγερμού. Πρόκειται για ένα σύστημα προειδοποίησης του Γιωργού εκείνου που κάνει λάθη, ούτω ώστε να αποφύγουμε μία απλή αφηρημάδα να μετατραπεί σε σοβαρή ποινή. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα για τους τίμιους γεωργούς που πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσω και το παράδειγμα το οποίο μας ανέφερε πολλές φορές ο συνάδελφος Ντες για το θέμα των ακουστικών που φόραγε στο δεξί αυτή ένας ε, γεωργός ε, και όχι στο αριστερό λέγοντας ότι έπρεπε να κοιτάει το, το, μοσχάρι του κατάπατσα. Πρέπει επίσης να σταθούμε και στην αναλογικότητα όπως επίσης για το θέμα της κύρωσης, δηλαδή το, να υπολογίζουμε και την καθυστέρηση και την πρόθεση. Για το θέμα των κυρώσεων να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο θα εμβαθύνουμε πολύ πιθανόν αύριο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τις κυρώσεις. Για το greening, το πρασίνισμα. Στις τροπολογίες εγώ τόνισα την ανάγκη να περιορίσουμε τις κυρώσεις αν έχουμε περιορισμένη εφαρμογή του greening μόνο στις πληρωμές του greening, του greening χωρίς ε, να υποσκάπτουμε την βασική πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί που δεν θα υποβληθούν στα μέτρα του greening θα πρέπει να χάσουν απλώς το μέτρο του greening και όχι την βασική πληρωμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί αυτή η ανάγκη για να μην έχουμε παρανοήσεις και δημιουργήσουμε τεράστιες δυσκολίες στους γεωργούς αυτήν την πρώτη φάση εφαρμογής της ΚΑΠ. Η προσπάθεια πλούστευσης θα πρέπει να εμπλέκει και τους γεωργούς και τα κράτη-μέλη, αλλά και τους οργανισμούς πληρωμιμών ή ελέγχου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα καθιστώντας το πιο ευέλικτο και μετρήσιμο ανάλογα με την απόδοσή του. Το κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει τον αριθμό των οργανισμών πληρωμής που θα έχει. Και αυτό ανάλογα και με το ρόλο δηλαδή που θα αναλάβει ο καθένας. Εγώ στην αρχή είχα προσανατολιστεί προς μια διαφορετική θέση. Εγώ ήθελα κάτι το πιο δεσμευτικό προς έναν ενιαίο ε, εθνικό οργανισμό πληρωμών. η διαφορετική διάρθρωση σε συναγματικό επίπεδο, συγκρότηση σε συναγματικό επίπεδο των κρατών μελών, οι διαφορετικές υπάρχουσες δομές ε, με έπεισαν για το αγαθόν της πρότασης της Κομισιόν. Ένα είναι σίγουρο ότι πέρα από τη συνταγματική διάρθρωση των κρατών μελών θα πρέπει ο βασικός στόχος των οργανισμών πληρωμών να είναι ο γεωργός και να του διασφαλίζονται ασφαλείς χρονικές στιγμές καταβολών πληρωμών. Δεν μπορεί ο Γιωργός να υφίσταται καθυστερήσεις γραφειοκρατικού ή άλλου τύπου. Εγώ σε τροπολογίες, στις τροπολογίες μου όρισα ορισμένα σημεία για να ορίσω την ακριβή ευθύνη όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και την υποδομή των διαφόρων χωρών στην εφαρμοστική φάση. Εγώ νομίζω ότι μία ανανεωμένη διαχείριση του συστήματος ελέγχου και, ταυτοπι... και διαπίστωσης ταυτοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των λαθών και των ελέγχων. Σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου, εγώ πρότεινα ορισμένες αλλαγές. Κατά πρώτον θα ήθελα να τονίσω το άρθρο 30 για την πρόταση για την ανάπτυξη της υπαίθρου που αναφέρεται στην δυνατότητα διπλής χρηματοδότησης και που αναφέρει αποκλειστικά τα μέτρα για τη βιολογική γεωργία. Εγώ ε, θέλησα να διευρύνω όλες τις αγροπεριβαλλοντολογικές πληρωμές του άρθρου 29 στην ίδια πρόταση, δηλαδή όλοι όσοι θα καρποθούν τον γεωργικό περιβαλλοντικών μέτρων θα τους αναγνωρίζεται αυτόνομα το greening δηλαδή αυτόματη αναγνώριση όχι μόνο για τη βιολογική γεωργία αλλά και για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τα όσα ψήφισε αυτό το κοινοβούλιο σχετικά με την προσαρμογή του οριζόντιου κανονισμού στην Λισαβόνα πρότισα η αυτόματη αποδέσμευση για τα προγράμματα της ανάπτυξης της υπαίθρου να γίνεται συνολικά από τα κράτη-μέλη και όχι μεμονωμένα. Ε, αυτό το συζητήσαμε πολλές φορές αυτή την Επιτροπή και το ενέταξα και στην τροποποιητική πρόταση του σχήματος της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εθνικές αντισταθμίσεις και στα κράτη-μέλη να πετύχουμε οι πιο δραστήριες περιοχές να μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια εκείνα τα οποία οι λιγότερο ικανές ε, περιφέρειες ε, δεν απορρόφησαν. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, ένα θέμα αντιμαχόμενο ε, το οποίο το συζήτησα και με τους άλλους εισηγητές αλλά δεν τα βρήκαμε. Πρέπει να το ξαναδούμε σε επίπεδο τροπολογιών και σε επίπεδο συμβιβασμών είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερους κανονισμούς και αφορά στην τοπική καινοτόμο συνεργασία. Εδώ δεν πρότεινα τίποτα. Θα το κάνω βεβαίως σε μια επόμενη φάση, διότι το να φαντάζεται κανείς ότι μπορούμε εμείς να παρουσιάσουμε προτάσεις σε τοπικό επίπεδο καινοτόμων σχεδίων που θα πρέπει να επιλεγούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο, μετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πολλά επίπεδα επαλήθευσης και ελέγχου για να χρηματοδοτήσουμε 50 προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα μάξιμο με 100.000 ευρώ. Ευρώ μου φαίνεται να είναι κάτι το πραγματικά ηλιγιώδες και σύνθετο με μικρές, ε, με μικρές επιπτώσεις. Νομίζω καλό θα ήταν να έχουμε μια ανταλλαγή best practice βελτιώνοντας τους ε, μηχανισμούς ε, για την ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών. Σχετικά με την, το ποσοστό προχρηματοδότησης των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, η πρότασή μου να πάμε στο 7% της ε, συμβολής του ΦΕΡΣΑ, οδηγεί σε μία στοχευμένη διαδικασία προγραμματισμού που θησαυρίζει την εμπειρία του παρελθόντος. Τώρα για τη νέα λειτουργία παρακολούθησης που εντάσσεται για πρώτη φορά θεωρώ ότι είναι θεμελιώδης όπως επίσης και η τυπολογία των κυρώσεων για να μπορέσουμε να πλουστεύσουμε τη ζωή των λειτουργών που θα έχουν ένα ενιαίο έγγραφο με τους δείκτες που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μετά το 2013 όπως επίσης εγκάρσια και τις παραβιάσεις. Θέλησα να διαγράψω την ε, εξουσιοδότηση προς την Κομισιόν, προτείνω καλύτερα δηλαδή τη διαγραφή της εξουσιοδότησης της προς την Κομισιόν για την ένταξη της οδηγίας για το νερό και για τα ζυζανιοκτώνα στη διαδικασία της αιρεσιμότητας. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτές οι θεματικές να αντιμετωπιστούν είτε με τακτική ad hoc διαδικασία είτε στο βασικό, στη βασική νομική πράξη να βάλουμε τα σημεία εκείνα τα οποία δεν θα μπορέσουν να είναι <coughs> αντικείμενο των διαφόρων εντεταλμένων πράξεων, εξουσιοδοτημένων πράξεων. Εγώ θα ήθελα να δούμε την πρώτη υπόθεση, να έχουμε δηλαδή μία ad hoc τακτική διαδικασία. Τελευταίο, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι όλες οι προτάσεις που διατυπώνουμε είναι προτάσεις ε, σχετικές ή συνδέονται με την πρόταση του MFF που διατύπωσε η Κομισιόν. Και έτσι όπως έχουμε γράψει όλοι οι συγητές, οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή της πρότασης του δημοσιονομικού πλευίου πλαισίου σε φάση ε, έγκρισης ε, θα χρειαζόταν διορθώσεις στις εκθέσεις μας. Πρότεινα ε, επίσης και μία σειρά αλλαγών με αναφορά στις έκτακτες συνθήκες γιατί μου φαινόταν περίεργο η Κομισιόν στην πρότασή της μεταξύ των διαφόρων ειδικών ε, περιστάσεων των ειδικών συνθήκων έχει διατυπώσει τις σχετικές επιζωτίες, τις επιδημίες των ζώων δηλαδή, χωρίς όμως να αναφέρεται στις φυτοπάθειες. Διότι ε, έτσι όπως τα ζώα μπορούν να αρρωστήσουν, αντίστοιχα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ασθένειες των φυτών. Επιτρέψτε μου τώρα να ολοκληρώνω ευχαριστώντας πρώτον τους εσκιώδεις εισηγητές, πιο συγκεκριμένα τον συνάδελφο Λάιον, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δυναμικός στις ε, προτάσεις του, όπως επίσης και όλους τους ε, παράγοντες της γραμματείας ε, των πολιτικών ομάδων που συνεργάστηκαν. Στην ομάδα εργασίας τη δικιά μου πρέπει να ευχαριστήσω τους βοηθούς της ομάδας μου που εργάστηκαν πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε όλες αυτές τις αλλαγές και τις τελικές προτάσεις στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Τζοβάνι. Σε ευχαριστώ και σένα για την εξαιρετική σου δουλειά. Πολύ σύνθετη δουλειά, πάρα πολύ <coughs> πολύπλοκη δουλειά. Και εδώ γράφτηκαν πολύ. Οπότε ρωτώ, παρακαλώ μάλλον συγγνώμη, να διαχειριστείτε όλοι καλά το χρόνο σας. Ο Ρέντσεκ και μετά George Λάιον. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον ε, εισηγητή μας που ετοίμασε αυτό το έγγραφο. Ε, η έκθεση αυτή προκύπτει από τα όσα θα δημιουργηθούν στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ακριβώς για αυτό το λόγο όλα αυτά θα τροποποιηθούν περαιτέρω, ανάλογα με το πότε θα ολοκληρώσουμε το έργο μας στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Αυτό αφορά και το greening, το πρασίνισμα και άλλα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη στάση εναντί του ελέγχου και του συστήματος άμεσων πληρωμών. Ό,τι τέλο πάντων καλύπτεται από το δεύτερο πυλώνα. Το έγγραφο αυτό σκοπό έχει να φροντίσει να υπάρχει διαφάνεια σε όλη του την έκταση. Δηλαδή, νική αρρωγή, στήριξη των γεωργών που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις άμεσες πληρωμές με διατάξεις που σίγουρα είναι βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες. Τώρα, ο έλεγχος και η παρακολούθηση και όλες οι ενέργειες της ε, ΚΑΤ με τρόπον ώστε να μην πληρώνουμε πολλά, να μην διασπαθίζονται τα κονδύλια, διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα χρήματα, για την περιουσία των κρατών μελών. Η διαχείριση της ΚΑΠ προποθέτει τεράστιες δαπάνες. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και αυστηρός ο έλεγχος, καθώς και η συγκράτηση του κόστους, όπου ο έλεγχος, μάλλον από τον έλεγχο, προκύψει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα λόγου χάρη των γεωργών. Εκεί ο έλεγχο μπορεί να περιοριστεί στα ερχόμενα χρόνια. Τώρα για τις κυρώσεις μετά από έλεγχο. Θα πρέπει να φροντίσουμε να τιμωρούνται μόνον οι γεωργοί που ενεργούν με διάθεση εξαπάτησης. Δηλαδή οι κυρώσεις να είναι ανάλογες με την συμπεριφορά των ε, γεωργών. Πρέπει μάλιστα να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ απάτης και απλού Οι φορείς πληρωμών είναι στοιχεία που θα πρέπει να... Ο τρόπος που θα λειτουργούν θα πρέπει να οριστούν από του ίδιου τους φορείς, δηλαδή η διαφάνεια, η ταχύτητα της ε, εκταμίευσης. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν ε, σε μία πρώτη φάση κατά αυτόν τον τρόπο για να σκεφτούμε μετά έναν ενιαίο φορέα. Όχι μόνο για να απλουστεύσουμε και να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά να ε, φροντίσουμε να καλύπτονται οι ανάγκε των γεωργών από αυτό το φορέα. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ και εδώ χρειάζονται διευκρινήσεις και βελτιώσεις. Έχουμε μια νέα δυνατότητα να δίνουμε να υποβάλλονται πολιετής μάλλον αιτήσει. Ένας γεωργός μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή άπαξ ανατριετία. Αυτό είναι μια λύση που την ζητούν ε, διακαώσει, οι Γεωργοί. Τα έγγραφα μπορεί να είναι εξαιρετικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και δουλειά μπροστά μας. Δηλαδή μετά τις εκθέσεις για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να ε, επανέλθουμε και να αποσαφενήσουμε το έγγραφό μας. Ευχαριστούμε ο κύριος, τον κύριο Ολενιτσακ και τώρα ο κύριος Λάιον. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας τον Τζοβάνι Λαβία για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με όλου του κοιόδης εισηγητές προσπαθώντα να βρούμε τι καλύτερε ιδέε και να βελτιώσουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του δημοσιονομικού και του οριζόντιου κανονισμού. Για πολλού. η μεταρρύθμιση αυτή τη ΚΑΠ αφορά τον πρώτο πυλώνα και τι άμεσε πληρωμέ. Όμω, η πραγματική ουσία τη μεταρρύθμιση επηρεάζει την καθημερινότητα των γεωργών ω προ τι κυρώσει τι ποινέ τους ελέγχους και πώς αυτά λειτουργούν. Έτσι, όπως ε, έχω δει να έχουμε από εκεί πολλά παράπονα, επιμένω πολύ στο συγκεκριμένο ντοσχέ, είναι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα. Και είναι ουσιαστική σημασία να προσπαθήσουμε να κάνουμε το σωστό. οι παρακολουθήσει, η πολλαπλή συμμόρφωση και οι κυρώσει να είναι λογικά σε σχέση με τον κίνδυνο που απομίζεται ο κάθε Γιώργος. Καλωσορίζω την θέση του Κοινοβουλίου που την έχει συμπεριλάβει ο ε, Τζοβάνι για τον ευθυγράμμιση. Αυτό είναι κάτι που ήταν απαραίτητο ώστε να μην αποδυναμωθεί η θέση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το πρόθεσμα. Υπάρχουν η κατεξουσιοδότηση πράξεις ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες και με αυτό θα προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν χρειαστεί. Έπειτα, η αρχή της προσέγγισης ανάλογα με τον κίνδυνο. Είναι σημαντικό που αυτό συμπεριλήφθη. Η μείωση του αριθμού των ελέγχων εκ των υστέρων εφόσον ένα σύστημα λειτουργεί εύρυθμα. Νομίζω ότι όταν κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του και αν μάλιστα οι αρχέ κάνουν τη ε, δουλειά του σωστά, οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να μπορεί να δίνει για κάποια επιβράβευση στους γεωργούς εφόσον ε, δεν κάνουν σφάλματα. Μείωση λοιπόν των ελέγχων είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Καλωσορίζω τα μέτρα για το greening, το πρασίνισμα και το μέγιστο των ποινών, των κυρώσεων και επίσης τις προτάσεις Καπούλα Σάντος. Το να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Εάν υπάρχουν αν υπάρχει σύστημα κυρώσεων, θα πρέπει και για τους γεωργούς που κάνουν σφάλματα τους δοθεί χρόνο ώστε να έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν τα σφάλματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διορθώνονται τα κακό και που υπάρχουν και όχι να επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Έπειτα η απλούστευση των αντίπων που έχει προταθεί και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό διότι οποιοδήποτε γεωργός δεν έχει αλλαγή στις συνθήκες όπου λειτουργεί ε, χρόνο το χρόνο είναι περίεργο να του και περιττό να του ζητάμε να συμπληρώνει ένα τεράστιο και τόσο μακροσκελέ έγγραφο κάθε χρονιά. Δηλαδή, τι να κάθεται ο άνθρωπο να γράφει φέτο ακριβώ όπω πέρσι. Χρειάζεται και χρόνο για να συμπληρώνεται αυτό. Οπότε όπου οι συνθήκες έχουν αλλάξει για τους γεωργούς, εκείνοι να συμπληρώνουν το ανάλογο έντυπο, αλλά ετησίως δεν χρειάζεται. Τελευταία παρατήρηση. Η ηλεκτρονική αναγνώριση ε, είναι μια σημαντική διάταξη όταν κανείς δεν μπορεί να τηρήσει πλήρως το μητρό για τα ζώα, θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει και μια ευελιξία να επιτρέπεται να διορθώσει την ε, καταγραφή. Εκεί που θα πρέπει να προσθεθούν κάποια στοιχεία είναι το κριτήριο για την υπολή των κυρώσεων θα πρέπει να υπάρχει ορισμό στη βασική νομίζω πράξη, διότι πολλά θα κρυθούν από αυτό. Έπειτα η αρχή για τις καταποκοπήν μειώσεις, αυτές θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση και εφόσον ισχύουν οι κυρώσει, θα πρέπει να είναι ο κίνδυνο για το Γενικό Ταμείο το κριτήριο. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αν έχουν συμπληρωθεί τα έντυπα όλα σωστά, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να επιβάλλεται μια κύρωση παρά όταν βλέπουμε αν υπήρχε ε, συμμόρφωση με τις απαιτήσει. Διότι ουσιαστικά η ουσία είναι ότι γίνεται με τον υπολογισμό της Επιτροπής και πώς αυτός πλήττεται, το γεωργικό ταμείο. Δηλαδή οι πολλές ζημιές, τα μικρά λάθη που έχουν γίνει εις βαρός αυτού του ταμείου θα πρέπει να είναι το κριτήριο η αρχή είναι να δούμε ποιο κίνδυνο μπορεί να ε, υπήρχε για το γεωργικό ταμείο. Αυτό ελπίζω να το συμπεριλάβουμε επίση στη βασική πράξη και να στηριχθεί. Δεν θα πω περισσότερα, διότι νομίζω ότι ο κύριος Λαβή έχει κάνει εξαιρετικό έργο. Ήταν ε, πολύ καλός συνεργάτης επίσης. Ήταν επικοδομητική η σχέση μας και νομίζω για τα δύο-τρία αυτά σημεία θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε. Ο Νίκολσον. <laughs> Συγγνώμη, Πρόεδρε. Άργησε η δίμηνια. Ναι, θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο Τζόρτζ και να ευχαριστήσω καταρχάς για, το, για την εξαιρετική έκθεση του εισηγητή. Πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένε εξαιρετικές ιδέες μέσα. Σίγουρα καλωσορίζω, ορισμένε προτάσεις. Είναι πολύ λογικές και πολύ συνετές. Αναφέρονται σε τομείς που θα διευκολύνουν την ζωή των αγροτών. διότι οι αγρότες είναι, έχουν μεγάλο φορτό εργασίας και η γραφειοκρατία επιβαρύνει τα πράγματα. Επίσης συμφωνώ σαφέστατα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, διότι πιστεύω ότι προς το παρόν είναι ένα σύστημα στινόμευσης παρά ένα σύστημα βοήθειας για τους ε, αγρότες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η κίτρινη κάρτα είναι μια καλή ιδέα ως έγκαιρη προειδοποίηση, ως επισήμανση του προβλήματος και η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών είμαι σίγουρος ότι με μια τέτοια κίτρινη κάρτα θα ασχοληθούν με την επίλυση του προβλήματος αυτού. Ε, επίσης πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε σε τοπικό σου περιφερειακό επίπεδο διότι προς το παρόν το κόστος, το διοικητικό κόστος είναι υψηλότατο, υπερβολικά υψηλό. Επίσης πιστεύω ότι είναι καλή η ιδέα να το αφαιρέσουμε αυτό από την πολλαπλή συμμόρφωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες. Η Κομισιόν αρνήθηκε να μας ακούσει όταν επισημάναμε τις αδυναμίες της CPID και πιστεύω ότι είναι πρέπον τώρα να μην δόθουν πινές στους αγρότες, να μην τιμωρηθούν οι αγρότες. Επίσης, όπως είπε και ο Τζόρτζ, πιστεύω πως μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά, αλλά τα βασικά είναι ήδη εδώ σε αυτή την έκθεση. Α μην επαναληφθώ. Α ευχαριστήσω ξανά τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά και ελπίζω να χτίσουμε πάνω στι γέρε βάσεις που έχει θέσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω την κελτική παρέμβαση τη συμμαχία που έχουμε κάνει εδώ. Σύμφων, ε, να συγχαρώ τον Τζιωβάνι, εξαιρετική δουλειά, πολύ δύσκολο το έργο, πολύ πλοκό. Ο δικός μας κοιόδης εισηγητής βρίσκεται στο Ρίο αυτή τη στιγμή, στέλνει τους χαιρετισμού του. Εγώ θέλω να συγχαρώ γενικά την έκθεση, αλλά ειδικότερα τις απλοποιήσεις θα μας δώσει κάποια ελπίδα ότι μπορούμε κάτι να καταφέρουμε, να δούμε ένα φως. Συγχαίρω επίσης τις αναφορές στις τεχνικές ε, αποτυχίες, στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις δυσκολίες που έχουμε στην εφαρμογή αυτών των ε, ταυτοποίησεων στους ε, κτηνοτρόφους προβάτων. Πολλά πράγματα λοιπόν είναι θετικά, οι απλοποίησει, η αναλογικότητα. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες βέβαια που στην εφαρμογή από τα επιμέρους Υπάρχουν πολλές διαφορές και δεν μπορούμε κατά ανάγκη εμείς να τα ρυθμίσουμε όλα από μία μόνο έκθεση. Ορισμένα σημεία που η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα ήθελε να δει πιο έντονα είναι η οροφή, εάν το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τις βιώσιμες αγροτικές πρακτικές, τότε θέλουμε να δούμε να χρησιμοποιηθεί αυτό για να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τη βιωσιμότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομιμότητα της ΚΑΠ Ας μην ξεχνάμε, πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Επίσης, θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο της παραγωγής τροφίμων. Προς το παρόν, στην Ευρώπη, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις είναι ολοένα και πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Θα θέλαμε λοιπόν να καλωσορίσουμε προτάσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το έδαφος, το νερό και επίσης να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για τις αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο για μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην υπάρχουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα για την οδηγία για το νερό, για, τα, για τη χρήση ζυζανιοκτώνων, για την χρήση των καταξουσιοδότηση πράξεων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα νομοθετικά όργανα που έχουμε και θέλουμε να δούμε να εφαρμοστούν το συντομότερο. Όταν έχουμε την ευκαιρία να, ε, να βελτιώσουμε κάτι, δεν πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Αυτά από μένα. Ο κύριος Ρούμπιξ. Ναι, ε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια λέει ο κύριος Σκοτά. Σημερίζομαι απόλυτα τις θέσεις ε, του συναντέλφου αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι ουσιαστικότατο για τη διαχείριση των ε, κονδυλίων στο κάθε κράτος μέλος. Οι τίτλοι 12 ως 15 της πρότασης για την χρηματοδότηση της διαχείρισης και παρακολούθησης της ΚΑΠ θα πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Συμφωνώ με τις τροπολογίες του κυρίου Λαβία για τον τρίτο τίτλο. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω το εξής. Για τους μελλοντικούς δικαιούχους της τεχνικής βοήθειας στη γεωργική εκμετάλλευση αλλά και για το κράτος μέλος που θα χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις το να οριστεί ένα ανώτατο όριο ε, τεχνικής ε, βοήθειας ε, το χρόνο ή αναδικαιούχο. Είναι ουσιαστικότατη η τεχνική βοήθεια για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς βεβαίως να χάνουμε από μπροστά μας και τους βασικούς ορίζοντες της κάποια. Να έχουμε αποτελε... Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφή και αποτελεσματική νομοθεσία σχετικά. Ευχαριστούμε κύριο Ρούμπεξ και μετά ο κύριος Ντέκ. Ευχαριστώ θεωρώ την έκθεση αυτή ενδιαφέρουσα. Καταγράφει μια πολύ καλή απεικόνηση για τα περισσότερα ζητήματα. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι τι γίνεται με τις άμεσες πληρωμές και την διάκριση των γεωργών που είναι ενεργοί ή όχι. Όταν επίσης καταγράφεται η έκταση μιας μονάδας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που είχαμε τον Ιούνιο του 2003, όμως οι συνθήκες μιας εκμετάλλευσης διαρκώς μεταβάλλονται μπορεί να υπάρχουν 150.000 εκτάρια περισσότερο από ό,τι είχαμε το 2003. Αυτό δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη, ακόμη. Ε, επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχει ανάγκη μεταβατικής περίοδου. Ίσως τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία ιδίως, να μην ε, συμμορφώνονται με τις, προ... με τις απαιτήσεις πλήρως αλλά θα πρέπει να τους δοθούν και άλλες επιλογές. Από το 2014 ίσως να υπάρχει δυνατότητα να ανατρέξουν και σε κάτι άλλο. Για τις ε, λιγότερο ευνεμένες περιοχές πρέπει να δούμε την απόσταση, τη μορφολογία, τη σύσταση του εδάφου ώστε μετά να φροντίσουμε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παρακολούθησα την έκθεση του κυρίου Λεβία με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον Ρούσα, η προσέγγιση του, οι αφετηρίες που χρησιμοποιεί, για την απαλληφή όσο το δυνατόν περισσότερο της γραφειοκρατίας, κάτι που σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο το ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά η γραφειοκρατία είναι κάτι που πρέπει να μειωθεί τώρα, να αναφερθώ στην εξαπάτηση, στην απάτη. Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους ελέγχους. Αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα σαφές όργανο. Τώρα όσον αφορά το greening θα ήθελα να δώσω την υποστήριξη της παράταξής μου σε εσένα, συνάδελφε Λαβία. Και να συμφωνήσω ότι χρειάζεται η πολλαπλή συμμόρφωση για να, εφαρμοστούν, για να εφαρμοστεί το greening, το πρασίνισμα. Για το χρηματοδοτικό πλαίσιο τώρα, επίσης σε υποστηρίζω, όμως μπορούμε να αποφασίσουμε καλύτερα όταν γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χρήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας και από πού. Και τότε μπορούμε να να, θα μπορέσουμε να ορίσουμε ποιος είναι ένας ενεργός αργότης, ποιος όχι. Τι γίνεται από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, γιατί όπως είπαμε το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Τώρα ο κανονισμός του 5% που αναφέρεται στην νομοθετική σας πρόταση δεν νομίζω ότι είναι, είναι καλό να παραμείνει. nie wiemy, jak to oceniają wyborcy. Pani poseł Jegle, następnie pani poseł Magines. Μάλιστα. Κύριε, κυρία Ιέγκλερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συναδελφό Λαβία. Πραγματικά η έκθεση είναι περιεκτικότατη, λεπτομερέστατη σε αυτή την έκθεση πραγματικά μπορούμε να δούμε πόσο σημαντική είναι η αποδόμηση της γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία έχει, είναι ένα πρόβλημα, έχει εγκατασταθεί και σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνατε προς την αποδόμησή της. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό και όχι και δεν θα ήθελα να ξύσω ανοιχτές πληγές εδώ τώρα για το πόσο θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι ή όχι. Σίγουρα δεν θέλουμε να ξοδέψουμε χρήματα των φορολογούμενων. Θέλουμε να τα ξοδέψουμε με όσο το δυνατόν πιο συνετό τρόπο. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε πολύ προσεκτικά ποιος, είναι ο στόχος και ποια είναι η γραφειοκρατία. Τι θα βλάψει αυτό τους στόχους μας γιατί όχι. Και εδώ αναφέρομαι στο θέμα των κυρώσεων. Είναι ο τομέας αυτός κάτι που απαιτεί πάρα πολύ εργασία, πάρα πολύ διοικητικό φόρτο. Θεωρώ πολύ σημαντικό και μάλιστα επαναλαμβάνεται η συμπερίληψη των περιβαλλοντικών μέτρων, το greening. Για μένα είναι σημαντικό να βρεθεί μία λύση η οποία θα αφορά και τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο εύκολο να λάβουν μια τέτοια πιστοποίηση από τις μικρές. Και σημαντικό είναι να δούμε τι θα γίνει με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις εφαρμοστικές πράξεις και να τις ελέγχουμε καλά. Είναι έργο μας ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. έχω μια παράκληση. Να κάνουμε τις έρευνές μας, να δούμε εάν δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι ή αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πότε, κάθε πέντε χρόνια, για παράδειγμα, να το αναθεωρούμε. Για και πώς θα γίνει αυτό, χρειαζόμαστε στατιστικές, χρειαζόμαστε πληροφορίες και χρειάζεται να καλλιεργήσουμε το σκεπτικό αυτό, να καλλιεργήσουμε την ε, ζήτηση στατιστικών στοιχείων, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε τις λύσεις τις οποίες αναζητούμε. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω και την έκθεση, γιατί πραγματικά έγινε μετά από μεγάλη συνεργασία και πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ επιτυχής και πρέπει να είναι και να είμαστε επιτυχείς. Κύριε Μαγκίνες, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Υποστηρίζω όλα του τα σχόλια σχετικά με το greening, με το πρασίνισμα και την αίτηση του να διαχωριστεί από τις ε, βασικές πληρωμές. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα που ξεχωρίζει τις κυρώσεις από τα λάθη. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μόνο σε μία συνεδρίαση. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν τα πάντα, πόση ακαμψία ή πόση ευελιξία υπάρχει στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μία συζήτηση επί της ουσίας και χρειαζόμαστε μία συζήτηση που να, βγάλει το, που να διαγράψει το αίσθημα φόβου στους αγρότες για τις κυρώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή, αυτή την προσέγγιση και ένα δίκαιο σύστημα λειτουργίας όσον αφορά για την Συμβουλευτική Επιτροπή των Αγροτών. Πραγματικά όλοι δεχόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα καλύτερο και πιο σβάθο σύστημα. Όμως μέσα στην, στα μέτρα λιτότητας που υιοθετούμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον ιδιωτικό τομέα που έχει για μένα ρόλο, μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο, όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις για το tagging. και για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των προβάτων. Εάν υπάρχει εκεί πρόβλημα στο σύστημα, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Και πραγματικά συμφωνώ ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στα λάθη. Και ίσως το φθινόπωρο μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό περισσότερο, να δούμε τι φταίει και το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Κύριε Βατσακόφσκι. Oh, Μάλιστα και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ, κυρία Ράιμερ έχει το λόγο, τον κύριο Λαβία για την εξαιρετική έκθεσή του. Ερώτηση, η πρόταση για να μην υπάρξει νέα τροπολογία αν δεν υπάρξει κάποια νέα, κάποιο νέο αίτημα. Ναι, το θεωρώ σωστό, όμως δεν θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις για παράδειγμα, των, ε, τις επιχειρήσεις που καλλιεργούν φρούτα, αν δεν υπάρξει νέος ορισμός, αν δεν υπάρξει διαχωρισμός ε, στο τι είναι καλλιεργήσιμη γη, τι δεν είναι. Για μένα, ό, οποιαδήποτε γη χρησιμοποιείται για να καλλιεργηθεί κάτι, ναι, είναι καλλιεργήσιμη γη. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτό δέντρο, φρούτο, λαχανικό, οτιδήποτε. Φυσικά και είναι αναγκαίο να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς και να δημιουργούνται εκ νέου καινούριε αιτήσει για χρηματοδοτήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε βήμα-βήμα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο εκ νέου. Να προσθέτουμε, να βρίσκουμε μία μικρή λύση, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, επιμέρους προβλήματα στις, στους παραγωγούς, στις εταιρείες αυτές. Γιατί με, τον σταδιακ... με τη σταδιακή αυτή αντιμετώπιση θα μπορέσουμε πραγματικά να τις βοηθήσουμε και δεν θα είμαστε στάσιμοι. Ας δούμε λοιπόν αν μπορούμε να βρούμε κάποια κάποια δυνατότητα για αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, βρίσκω εξαιρετική την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βοητσακόφσκι. Ευχαριστώ. Όταν μίλησε η κυρία Γέγκλα για τις στατιστικές, θυμήθηκα Κάτι που έλεγε ο Γιούλιαν Τούβιμ, ένας Πολωνός του 19ου αιώνα. Έλεγε ότι υπάρχουν τριών ειδών ψέματα. Το σύνηθες ψέμα, το λευκό και μετά το στατιστικό. Άρα και στην Πολωνία, όπως και σε άλλες χώρες, οι, Πολωνοί, οι Γεωργοί έχουν πολλά προβλήματα. και με τις διάφορες υπηρεσίες και βεβαίως με το πώς μπορεί να υπολογίζονται οι κυρώσεις τους λόγω των σφαλμάτων μπορεί να έχουν γίνει, όμως αυτά τα επομίζονται κυρίως οι χειοργοί. Ένα σφάλμα ακόμη και αφελές ενός γεωργού μπορεί να γίνει και να μετατραπεί σε απάτη. Ε, στην Πολωνία λοιπόν έχουμε χιλιάδες εγκληματίες από αυτή την έννοια. Δεν μιλάμε όμως εδώ ούτε για εξαπάτηση ούτε για εγκληματίες στην πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά τιμωρούνται δύο φορές. Πρώτον γιατί τους ε, ανακαλείται η πληρωμή και δεύτερον διότι κρίνονται από τα δικαστήρια για ε, υποθετικές καταχρήσεις. Έτσι λοιπόν ε, είναι σημαντικό που ο εισηγητής μας έλαβε υπόψη και αυτό το, αυτή τη διάσταση. Για γραφειοκρατικούς λόγους οι γεωργοί δεν μπορεί να ε, υφίστανται όλα αυτά που σήμερα τους ε, αναγκάζουν να υποστούν. Θα πρέπει αυτό το σύστημα κυρώσεων υπερβολικών κυρώσεων να παλευθεί. Θα πρέπει οι κυρώσεις κατά των γεωργών να επιβάλλονται μόνο εφόσον υπήρξε σφάλμα ε, σοβαρό και όχι μια απλή απλεψία Και μια καθοριστική παρατήρηση νομίζω. Ε, η επόμενη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή που το έλαβε υπόψη. Τώρα και σε μια από τις προηγούμενες εκθέσεις μας, όπως ε, την έκθεση Σρόιτερ που μιλούσαμε για απλούσταση της ΚΑΠ και σε εκείνη, το πρόβλημα αυτό είχε ήδη εντοπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε ώστε οι γεωργοί να μην είναι θύματα των ε, κυρώσεων. Σας ευχαριστούμε μίλησε ο πρώην ε, εισαγγελέα και πρώην δικαστής ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και τώρα ο κ. Καπουλάς Σάντους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ προφανώς να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Λαβία για τη δουλειά του και για την μέρημνά του να διαδρώσει θέσεις με όλους τους συναδέλφους, ιδίως τους υπόλοιπους εισηγητές. Έτσι, η κοινή μας δουλειά μπορεί να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και συνένεση. Η δουλειά του δεν ήταν απλή. Υποβλήθηκαν προτάσεις που πρέπει να συμφιλιώσουν την απλούστευση που όλοι επιζητούμε με την απαραίτητη αυστηρότητα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στους πολίτες να διαφανεί ότι Θέλουμε να τους διευκολύνουμε και όχι να είμαστε αυστηροί με δημόσιο χρήμα, δημόσιους ελέγχους. Εδώ θα πρέπει όλα αυτά να ασκούνται με πλήρη συνέστηση και αυστηρότητα. Μιλάμε λοιπόν για μια έκθεση ιδιαίτερα περίπλοκη από τεχνική άποψη. Ακριβώ γι' αυτό εκτιμώ ακόμη περισσότερο τη δουλειά του συναδέλφου και να επιστήσω την προσοχή σε δύο σημεία. Δύο σημεία που έχουν να κάνουν με πράγματα που θα τα συζητήσουμε έτσι αλλιώ και αύριο. Πρώτα απ' όλα, το τι γίνεται με τις ε, μεμονωμένες κυρώσεις για τις βασικές πληρωμές και για τις πληρωμές πρασινίσματος, Εδώ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εισάγουμε έναν μηχανισμό που να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση ο παραβάτης να μπορεί να δικαιούται ε, ωφελών ε, χάρη στην παράβασή του. Αυτήν την διευκρίνηση πρέπει να την κάνουμε διότι μπορεί να προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι αυτό της διπλής χρηματοδότησης. Θα μου προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ε, διατηρήσει το άρθρο 30 που έχει εισάγει. Εκεί μιλά για την εξαίρεση της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των μέτρων ε, βιολογικής ε, γεωργίας του δεύτερου πυλώνα και του greening. Ενώ ο εισηγητής πολύ σωστά κάνει και επικροτεύω την ε, επιλογή του, διότι πραγματικά λαμβάνει υπόψη τη δική μου την πρόταση. Εδώ λοιπόν προτείνει την ίδια μεταχείριση για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτά και εγώ θα έλεγα ότι λογικό θα ήταν να συμπεριλαμβάνονται ως αντίστοιχα ισοδύναμα του greening. Όμω, το άρθρο αυτό καθεαυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι η ύπαρξη τέτοιο άρθρο στον κανονισμό ουσιαστικά μα αναγκάζει να παραδεχτούμε ή τουλάχιστον υπονοεί ότι υπάρχει διπλή πληρωμή. Κάτι που δεν ισχύει, διότι σε αυτή τη φάση, όπω γνωρίζετε, Κάποιες, κάποιοι από τους ισχύοντε ε, κανονισμούς επιτρέπουν άμεσες πληρωμές, αλλά για τις ίδιες επιφάνειες. Ε, πληρωμές για την ε, βιολογική γεωργία και για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Όπως ξέρετε, δεν γίνεται θέμα διπλής πληρωμής εκεί. Για τον επιπλέον λόγο, και θα το δούμε αυτό και στον κανονισμό για την ανάπτυξη της Πέθρου, για τον επιπλέον λόγο ότι όλα τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα πρέπει να είναι πρασινότερα, απαιτητικότερα από την πλευρά την περιβαλλοντική σε σχέση με τα μέτρα που προτείνονται για το greening. Η βιολογική γεωργία μάλιστα περισσότερα από όλα τα άλλα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα αφού είναι το αγροπεριβαλλοντικότερο όλων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσον μπορούν αυτά τα δύο ζητήματα να εξαιρούνται ή αν απλώς πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 30. Μήπως αυτή η αν Μα πρεπει να διαγραφει το αρθρο 30 μηπως αυτη η διαγραφη μα οδηγεί στο να παραδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση διπλής χρηματοδότησης, διπλής πληρωμής. Ο κύριος Ντότς. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, καλωσορίζω και εγώ την έκθεση. Εμείς ως Ευρωβουλευτές πιστεύω πως ξοδεύουμε πολύ χρόνο μιλώντας για απλοποιήσεις, λες και είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, λες και είναι κάτι που ποτέ δεν καταφέρνουμε. Όμως χαίρομαι γιατί δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό, αλλά τώρα έχουμε και κάποιες ιδέες για το πώς θα γίνει αυτή η απλοποίηση και πώς θα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ υποστηρίζω έντονα την απλοποίηση. Όταν πηγαίνω στην εκλογική μου περιφέρεια σε συναντήσεις αγροτών, πάντα προκύπτει κάποιο σχετικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η πρόταση είναι εξαιρετική για τις απλοποίησεις. Επίσης το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που δίνει στους αγρότες τη δυνατότητα να διορθώσουν τα λάθη τους. Οι αναφορές στα, στις ποινές καταποκοπήν και στην πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό το όργανο είναι κάπως χοντροκομμένο, δεν είναι αναλογικό. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να το να αναλογιστούμε περισσότερο πώς θα διαφοροποιήσουμε την απάτη, την εσκεμμένη απάτη και το λάθος. Διότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο οικονομικών δυσκολιών και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το πώς ξοδεύουμε το δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι πάλι και οι ίδιες αρχές που αναφέρονται στην πολλαπλή συμμόρφωση υπάρχουν και εδώ και χαίρομαι που θα τις κοιτάξουμε σε εθνικό επίπεδο. Χαίρομαι επίσης που ορισμέ... πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη χρησιμοποίησαν το καταποκοπήν σύστημα κυρώσεων. Και στη Βόρεια Ιρλανδία η δική μου εμπειρία έχει, μου έχει διδάξει ότι αυτό είναι δυσανάλο... δυσανάλογο με τον πραγματικό κίνδυνο και το σύστημα αυτό έχει οδηγήσει σε προβλήματα για τους αγρότες. Όταν λοιπόν εξετάσουμε την απλοποίηση πρέπει να το κοιτάξουμε. Σε γενικές γραμμές όμως είναι εξαιρετική η έκθεση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την κατεύθυνση την οποία παίρνει και για τις τροπολογίες θα σκεφτούμε και θα σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Ευχαριστούμε, κυρία Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαβία. Πραγματικά ασχολείται ενεργά για την ε, αποδόμηση της γραφειοκρατίας και είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αγρότες όσον αφορά τον κατάλογο των κυρώσεων. Πιστεύω ότι ε, συμφωνώ με όσα είπε η προλαλή σας. Στη Γερμανία υπάρχει ε, ένα καταποκοπήν ε, ποσό και η πληρωμή είναι η ίδια για οποιαδήποτε έκταση. Γενικά υπάρχει ε, πρόβλημα δυσαναλογίας. Και για μένα είναι πολύ σημαντικός ο διαχωρισμός όταν μιλάμε για κυρώσεις. Ή λάθη και πώς μπορούμε να διορθώσουμε ένα λάθος και πότε αυτό είναι λάθος. Και πότε ένα λάθος δεν διορθώνεται. Μετά για την πολιετή έκθεση. Η συνάδελφος Γέγκλερ ήδη το ανέφερε. Είμαστε ίσως λίγο υπερβολικά αισιόδοξοι. Σε εμάς τη Γερμανία δεν αποτελεί αυτό πρόβλημα. Υπήρξε και στο παρελθόν ε, ηλεκτρονική πρόσβαση. Το καταφέραμε βέβαια με πολύ κόπο αυτό να αποκτήσουμε δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά, για παράδειγμα στο, στην καλλιέργεια των σιτηρών, του κρυθαριού. Το σημαντικό για μένα δεν είναι η αιτήσει αναέτος, αλλά ο έλεγχος που θα πρέπει να γίνει στις αιτήσει αυτές, όχι ο αριθμός τους. Μετά, εξαιρετική ιδέα για τις ε, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα και για το πρασίνισμα και για την, απελευθε... Ε, για την απελευθέρωσή τους από την υποχρέωση πρασινίσματος. Και είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να φτάσουν σε αυτόν τον στόχο. Να τις διευκολύνουμε. Μετά. Όσον αφορά το no money no vote. Τα χρήματα, τα κονδύλια. Όντως ο προπολογισμό μας είναι πολύ μικρότερος και πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να πω ότι δεν κατανέμονται δίκαια τα κονδύλια. Είδαμε για παράδειγμα την περίπτωση των προβάτων και, των, ε, και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Δεν μπορώ πάντω εγώ να φανταστώ ότι για τα πρόβατα, για παράδειγμα, πρέπει να ισχύσουν διαφορετικοί κανόνες ταυτοποίηση για τα, παρά για τα βοηδή. Ευχαριστούμε κυρία Καλνιέτε. Ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω την έκθεση του κυρίου Λαβία. Η έκθεση αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και πραγματικά έχετε όλο το σεβασμό μου, κυρία Λαβία. Στην δική μου χώρα, στη Λετωνία, υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός για το, ανάμεσα στο πρασίνισμα, στις άμεσες ενισχύσεις, στους αγρότες. η προϋποθέσεις για αιτήσει άμεσων πληρωμών είναι αρκετά περίπλοκες. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να έχαναν οι αγρότες όλες αυτές τις άμεσες πληρωμές με... χρησιμοποιώντας αυτήν την διαδικασία. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα δύσκολα σημεία. Παράγραφος 8. Οι απαιτήσει για τις πληρωμές, για την οργάνωση των πληρωμών, αυτό θα πρέπει για μένα, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά τη γνώμη μου τις κατεξουσιοδότηση Τα κράτη-μέλη θα, θα πρέπει για μένα να διαχωριστούν από, σε αυτή τη διαδικασία. είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας και να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Εμείς έχουμε λοιπόν τις αμφιβολίες μας για τη χρήση των κατεξουσιοδότησης πράξεων. Πιστεύουμε ότι αυτό θα επιβάρυνε τα κράτη-μέλη. Επίσης, έχουμε ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά τον έλεγχο για τα ιδρύματα πιστοποίησης. Ανησυχούμε ότι αυτό θα προσθέσει επιπλέον διοικητικό φόρτο και επιπλέον κόστος και θα κάνει τη ζωή των αγροτών πολύ πιο δύσκολη. Να ευχαριστήσω τέλος τον εισηγητή για την πρόταση που διατύπωσε στο άρθρο 34 για την αλλαγή της ε, πρότασης χρηματοδότησης στο 7%. Για μας είναι σημαντικό αυτό. Και θα επανέλθω με τις προτάσεις μου ως τροπολογίες. Ευχαριστούμε ο Ροχάσινικ. Ροχάσνικ. Μάλιστα, πρέπει να εξετάσω τις, όλες αυτές τις προτάσεις. Για τους ελέγχους όμως να πω ότι εμείς ε, χρησιμοποιούμε το σύστημα των ε, βέλτιστων πρακτικών και αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι αποδοτικό, δουλεύει το σύστημα. Άμα ναι, να δούμε πώς θα το μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πολλά κράτη-μέλη είμαι σίγουρο ότι το, το, το σύστημα που χρησιμοποιούν δεν είναι αποδοτικό. Όμως θα ήθελα να πω τώρα κάτι που αντιτίθεται σε αυτά που είπε ο Πίτερ. Ότι όλα τα περιβαλλοντικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που, σκε... που θα εξισώνονται με την βιολογική γεωργία όσον αφορά το greening. Εκεί διαφωνώ. Έχουμε κάποια μέτρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ όμως να πω για όλα αυτά ότι κάθε πρότυπο θα πρέπει θα αναγνωρίζεται ως φιλικό προς το περιβάλλον. Στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά στάνταρ και διαφορετικά πρότυπα για την οικολογική γεωργία. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διαφωνήσω με την κοινή αυτή η θεώρηση. Δεν μπορούμε, δεν είναι όλα ίδια, δεν μπορούμε να τα, θεωρήσουμε, να τα αξιολογήσουμε όλα με τον ίδιο τρόπο. Γενικά όμως συμφωνώ με τα υπόλοιπα. Krótko pani Jeglen, rozumiem, że jakieś wyjaśnienie, sprostowanie. Mamy chwilę czasu. Μάλιστα. Τώρα, πριν ήταν Ιρλανδοί, τώρα συζητούμε μεταξύ μας τα γερμανικά. Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά μέτρα νομικά μέτρα. Όταν, όταν χρησιμοποιούμε μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν, τα οποία έχουν νομική βάση, τότε πραγματικά πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες, πραγματικά θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση, πραγματικά θα έχουμε καλές βάσεις και θα μπορέσω να υποστηρίξω και την πρόταση Λαβία. Πρέπει όμως να μην, μιλάμε θεωρητικά, πρέπει να, δούμε, να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Με τα λόγια πολλά γίνονται. E, Ευχαριστούμε. Και τώρα ο Διευθυντής Πατσέκο. Jaka musi być skala, wielkość programu prośrodowiskowego, aby być uznanym... Αλλά ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Ποιο θα, είναι το, θα πρέπει να είναι το, η έκταση ενός ε, προγράμματος βιολογικού για να καλύπτει τις προϋποθέσεις του greening. Διότι από, αυτό που, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ θα πρέπει κάποιο να είναι μετρήσιμο αυτό το μέγεθος. Έπειτα για τις κυρώσεις. Στο 30% των πληρωμών. Εάν δεν υπάρχει greening, η κύρωση φτάνει το 30% ενώ αν κάποιος γεωργός είναι τελείως ε, αντιορθόδοξο στην παραγωγή του. Παράγοντας λόγω χάρη Δημητριακά, τι θα πούνε οι, οι εμπειρογνώμονες. Δεν θα ασκήσουν κριτική. Διότι εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, όμως κατά πάσα πιθανότητα οι πιο πράσινοι εντό εισαγωγικών θα τηρήσουν διαφορετική στάση. Και το τρίτο στοιχείο, Το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και πληροφόρησης. Ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι γεωργοί, όπως και άλλες κοινωνικές κατηγορίες, δεν συμμορφώνονται πάντοτε με όλε τι προποθέσει. Πάντοτε θα υπάρχει κάποιο κάποιος που κάτι δεν κάνει σωστά, λόγω χάρη με τη χρήση των ε, ή με, την, τα, με τα πρότυπα παραγωγή τροφίμων. Θα χρειαζόταν λοιπόν ενδεχομένω μεγαλύτερη αυστηρότητα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <coughs> θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Λαβία για την έκθεσή του. Είναι πολύ αναλυτική, πολύ εμβαθυμένη και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί του επικοδομητικά. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την υποστήριξή του στις προτάσεις της Κομισιόν για τους οργανισμούς πληρωμών, όπως επίσης πιστεύω ότι πολλές από τις τροπολογίες που προτάθηκαν όπως επίσης και πολλά από όσα υπόθηκαν από πολλούς βουλευτές σήμερα τίνει προς την κατεύθυνση των θέσεων της Κομισιόν. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο γεγονός της προσαρμογής των ελέγχων όταν διαπιστώνουμε μικρά λάθη ή το πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε τα αιτήματα των ε, γεωργών, ας πούμε, να έχουμε ερωτηματολόγια προσυμπληρωμένα, για παράδειγμα, σε επίπεδο κρατών μελών. Θα ήθελα επί όμως, παρόλα αυτά, να εκφράσω την αντίρρησή μου για συγκεκριμένα σημεία. Πρώτο, ζητείτε να αναχθεί σε εθνικό επίπεδο ο κανόνας M2 αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα, διότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά στο στρατηγικό πλαίσιο, που δεν αφορά μόνο στις δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου, αλλά και σε άλλα διαρθρωτικά ταμεία. Μας δημιουργεί πρόβλημα λοιπόν. <coughs> Ένα άλλο θέμα, το οποίο έθεσαν και άλλοι βουλευτές, είναι το θέμα των κυρώσεων σχετικά με το greening. Άκουσα αυτό το οποίο υπόθηκε διάβασα αυτό το οποίο προτείνει ο εισηγητής. Αλλά έχουμε εδώ ένα πρόβλημα, ένα σημαντικό πρόβλημα. Εάν εμείς ακολουθήσουμε αυτό που μας λέτε, δηλαδή οι κυρώσεις για το greening περιοριστούν στο όριο που, στο ποσό το οποίο ανήκει το greening, εμπίπτει στο greening, τότε τι σημαίνει αυτό, ότι το greening αποτελεί προαίρεση. Δηλαδή άμα δεν θέλει ο καλλιεργητής το greening τότε δεν παίρνει τη βοήθεια. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι ένα μέτρο όπου το greening, το πρασίνισμα θα βρίσκεται στο επίκεντρο των αμέσων πληρωμών και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις. Και αν οι κυρώσεις μπορούν να ξεπερνάνε την ενίσχυση δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να κάνουμε εξαίρεση για το greening. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι η καταβολή των προκαταβολών. Εδώ έχουμε ένα θέμα διαχείρισης, δημοσιονομικής διαχείρισης. Αν εμείς επιτρέπαμε την καταβολή των προκαταβολών πριν από τις 16 Οκτωβρίου, αυτές θα πληρωνόντουσαν από τον προϋπολογισμό του προηγουμένου οικονομικού έτους. Και εδώ θα δημιουργούσαμε προβλήματα διαχείρισης του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό. Επιστήνω την προσοχή σας λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο αλλά σημαντικό σημείο. Άλλο, συμπερίληψη της οδηγίας πλαίσιο για το νερό και για τη χρήση των ζυζανιοκτώνων στην αιρεσιμότητα. Ε, θα ήθελα να δώσω ένα σαφές μήνυμα εδώ. Πρόκειται για οδηγίες πολύ σημαντικές. Αλλά αυτές οι οδηγίες γίνονται έχουν υπόσταση όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και αυτό ορίζεται στον κανονισμό. Για την ευθυγράμμιση με, με τη Λισαμπόνα πρόκειται για ένα οριζόντιο ζήτημα το Κοινοβούλιο επίσης θα λάβει οριζοντίως θέση. Πρόκειται για ένα θέμα το, για το οποίο θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Και παρουσιάσαμε συμβιβαστικές προτάσεις σχετικά. Για ένα ειδικό θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Η ηλεκτρονική ταυτότητα για τα κατσικοπρόβατα αυτό δεν εντάσσεται στην αιρεσιμότητα. Αλλά στο γεγονός ότι στον κανονισμό 21 του 2004 που είναι ο βασικός κανονισμός κάτι τέτοιο προβλέπεται. Δεν ε, αλλάζοντας κάτι τέτοιο στον τωρινό κανονισμό δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα το πρόβλημα, εάν υπάρχει, βρίσκεται στον κανονισμό, στον βασικό κανονισμό των 21 του 2004. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Διευθυντά. Παρακαλώ τώρα τον εισηγητή να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλες τις χρήσιμες προτάσεις που υπέβαλαν και που <coughs> διαπάνηκαν και κατά τη συζήτηση. Θα βελτιώσουμε λοιπόν τη δουλειά μας. Πάντα ε, διαπιστώνω ότι υπάρχει συνένεση σε πολλά θέματα όπως είναι η απλούστευση, η μείωση της, του γραφειοκρατικού άχθους για τους ε, γεωργούς, υπάρχει συνένεση για το θέμα της ε, έγκαιρης προειδοποίησης, ε, δυνατότητα, ε, μια που είμαστε και σε περίοδο ποδοσφαιρική, συμφωνία για αυτήν την κίτρινη κάρτα που θα πρέπει να δίνουμε στο Γιωργό ο οποίος κάνει μικρό Έχουμε ακόμη πολλά να συζητήσουμε βέβαια. Ετέθησαν ερωτήσεις από, από συναδέλφους και είναι υποχρέωσή μου να απαντήσω. Λέω στον συνάδελφο έχω τη σαφώς και λείπει ο ορισμός του τι εστί ενεργός γεωργός, διότι αυτός ο κανονισμός αποτελεί κομμάτι ενός πακέτου. Και αύριο θα δούμε τι θα μας παρουσιάσει ο συνάδελφος Κάρλος Σάντος με την αναφορά στις άμεσες πληρωμές. Και φυσικά γύρω από όλα αυτά εμείς θα πρέπει να διασυνδέσουμε όλες τις προτάσεις. Το γεγονός ότι έχουμε τέσσερις ε, κανονισμούς μας επιβάλλει να, να συμβρεθούμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για την καινοτομία. Εγώ δεν είμαι σαφής σαφώς υπέρ αλλά για την συνεργασία, την καινοτόμα συνεργασία, για τον οριζόντιο κανονισμό, για τη χρηματοδότηση κτλ. Αυτό θα προκύψει από το τι θα αποφασίσουμε στον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αν εμείς αυτόν τον κανονισμό αποφασίσουμε κάτι για την καινοτόμο συνεργασία κλπ τότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τις υπόλοιπες εκθέσεις χρειάζεται δηλαδή εμείς να κάνουμε μία συναρμολόγηση στο τέλος ένα θέμα το οποίο μου φάνηκε εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της απλούστευσης με τις ε, πολυετές με τις πολιετής αιτήσει. Αυτό για να αποφύγουμε. Γεωργοί που έχουν μία γεωργική εκμετάλλευση σταθερή και μία επιχειρησιακή μορφή σταθερή, να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να υποβάλουν την ίδια αίτηση. Η κυρία Ράιμερς η οποία έφυγε έλεγε Μα αν άλλαζε η δομή της ε, γεωργικής εκμετάλλευσης, τι γίνεται με μία ας πούμε επέκταση Μα φυσικά τότε αλλάζει η δομή και τότε γίνεται και η αντίστοιχη προσαρμογή στην έτσι. Εξ, επίσης θεωρώ απαραίτητο πέρα από την απλούστευση να υπάρξει και σχετική προσοχή και αυστηρότητα ε, δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε δημόσιο χρήμα στις προτάσεις ε, που κάνουμε. Ο ρόλος για την ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών πιστοποίησης τίνει στο να τίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να μειώσουμε το άχθος για τους γεωργούς μετατοπίζοντας το θέμα του ελέγχου και των επαληθεύσεων σε άλλο επίπεδο. Αν αυτό για τα κράτη-μέλη σημαίνει κάποια διοικητική δαπάνη επιπλέον, συμβάλλει όμως στο στόχο που εμείς θέσαμε αυτούς, δηλαδή την απλούστευση της ζωής των γεωργών, διατηρώντας και το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου. Επίσης ο συνάδελφος Κάπουλας αναφερέθηκε στο άρθρο για τη διπλή χρηματοδότηση. Αν δεν θυμάμαι καλά στην ανάπτυξη της υπαίθρου μιλάμε για τις αγροπεριβαλλοντικές επιπτώσεις στο κέρδος και στα, στις δαπάνες που προκαλούνται από την οικοαϊφορία. Μα για τον ίδιο λόγο θα πληρώνουμε εμείς και από τις δύο μεριές. Δηλαδή άμεσες πληρωμές από τη μια και από την άλλη μία αποζημίωση για το κόστος. Σωστά έλεγε ο συνάδελφος Σικέρσκι ότι η κύρωση για το 30% του greening την χάνει ορισμένων κριτικών για, για αυτούς που είναι πιο ευαίσθητοι για τις θεματικές προβληματικές. Όρι, κάποιος από εδώ πρότεινε, στην Επιτροπή μας δηλαδή, η κύρωση για το greening να ξεπερνάει και την ε, βασική πληρωμή. Θα τα συζητήσουμε αυτά όμως. Για το θέμα που έθεσε ο Διευθυντής Πατσέκο. Το θέμα των commitment σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή εφαρμογή του, M, ε, του M2 σε εθνικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο το Κοινοβούλιο μας το έθεσε συγκεκριμένα ως προς την ευθυγράμμιση και ψηφίστηκε σε αυτήν την Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Οπότε θεώρησα σωστό να το βάλω στην έκθεσή μου. Εγώ τότε το είχα καταθέσει ως τροπολογία και το ξανάφερα. Μπορεί να δημιουργεί μπερδέματα, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε δίκαιοι με τα κράτη-μέλη. Εντάξει υπάρχουν κράτη τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά από ό,τι άλλο, οπότε εδώ ίσως την κατάσταση. Είναι σαφές ότι η κύρωση περιορισμένη για το 30% στο greening ε, de facto οδηγεί το greening στην προαιρετικότητα, μα αυτή είναι μια επιλογή. Δεν είναι μια θέση, είναι ε, τυχαία, είναι σαφής επιλογή. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή μας, το συζητήσαμε και οι εισηγητές και αυτή είναι η πρότασή μας. Πιστεύω όμως, ή τέλος πάντων στην ερμηνεία μας ήταν διαφορετικό το θέμα των προκαταβολών. Εμείς για τις 16 Οκτωβρίου δηλαδή, για τις άμεσες πληρωμές, ήταν για ειδικέ καταστάσεις. Έτσι συνέβη στο παρελθόν δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά τι έγινε στην Ιταλία με τον σεισμό στη Λάκουιλα ζητήθηκε και παραχωρήθηκε διότι υπήρχε φυσικά και το κονδύλι η προκαταβολή. Ήταν αυτή η βούληση του να διατηρήσουμε ένα ζήτημα δυνατο, ανοιχτών δυνατοτήτων για να μπορούμε δηλαδή να χορηγούμε προκαταβολές. Εγώ καταλαβαίνω ότι σε συστηματική εφαρμογή θα είχαμε το πρόβλημα του οικονομικού έτους. 15 Οκτωβρίου κλείνει το οικονομικό έτος σε γεωργικό επίπεδο, θα δημιουργούσε λοιπόν προβλήματα στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Για το θέμα της ερεσιμότητας, για την οδηγία, για το νερό και για τα ζαρνιοκτώνα, θέλουμε να συζητήσουμε αναλυτικά τα περιεχόμενα και όχι να τα συμπεριλάβουμε. Σίγουρα όμως έχουμε χρόνο γι' αυτά. Τελευταίο, το χρωστάω, γιατί προηγουμένως δεν το έκανα. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τις υπηρεσίες της για, τις, για τη συνεργασία. Γιατί στα πλαίσια της διαδικασίας μας βοήθησε και πρέπει να την ευχαριστήσουμε. σε πολλές περιπτώσεις όπως το θέμα του οργανισμού πληρωμών βέβαια πολύ από τη δουλειά την αφήσαμε παράμερα γιατί χρειάστηκε να κάνουμε άλλου είδους πολιτικές επιλογές περιμένω και άλλες προτάσεις για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε όλο μας το έργο και να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα συνάδελφοι φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασης 9 Ιουλίου το μεσημέρι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές ε, για, την, ε, για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Είχαμε μία συζήτηση πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ ενεργή. Πολλοί μίλησαν τρεις φορές. Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ καλά τη βδομάδα μας. Στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί.